Ε, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ καθίστε. Ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ε, σας έχουμε ενημερώσει για την ακύρωση του σημείου 5 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση κλέβα και ακούς πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Έχει κυρωθεί επίσης και το σημείο 6, πρόληψη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη μομοποίηση εισόδων παράνομες δραστηριότητες. Κάρεν είναι ο εισηγητής. Και για το σημείο 10 προβλέπεται μία αναβολή βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα. Έκθεση Μπέρες. Να συμπενθυμίσω επίση ότι αύριο θα ξεκινήσουμε στι 10 το πρωί με μια ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα κάνουμε και κάποιες ανακοινώσει αφού προηγηθεί η ανταλλαγή απόψη, απόψεων με τον Επίτροπο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αύριο στις 10 το πρωί. Η ανταλλαγή απόψεων όμως με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα γίνει το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 4.30 και θα συνεχίσουμε μετά τις 4.30 με τα υπόλοιπα θέματα της Επιτροπής μας. Θα ήθελα λοιπόν ευθύ αμέσω να καλωσορίσω τον Επίτροπό μας. Όπως πάντα είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μας και χαρά για μας να ανταλλάσσουμε απόψει ε, για τις πρόσφατες εξελίξεις ε, όσον αφορά την ενιαία αγορά. Επίση ήσασταν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ, επομένω μπορεί να μα πείτε περισσότερα πράγματα όσον αφορά το μηχανισμό ESM την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους και χρηματοδότησης ε, κρατών εκτός Ευρωζώνης, όπως Νομένο Βασίλειο για παράδειγμα, και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να έχουμε σήμερα την ανταλλαγή αυτή απόψεων, γιατί βρισκόμαστε μία μέρα μετά την επέτειο της κρίσης ε, της Lehman Brothers, θα ήθελα λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε λίγο όσον αφορά την κοινοτική νομοθεσία. Επίση, σήμερα το πρωί υπάρχουν πάρα πολλέ εφημερίδε οι οποίε ε, αναφέρονται σε πρώην ε, διοικητέ τραπεζών όπω ο κύριο Ντάμον από την Barclays, ο οποίο λέει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη τυποποίηση και προστασία των καταναλωτών και των αγορών και ότι δεν μπορούμε πλέον να προχωρούμε περισσότερο με το λογότυπο too big to fail, ότι κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά για να καταρρεύσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ ισχυρή νομοθεσία όσον αφορά την χρηματοπιστωτική νομοθεσία και την ενιαία αγορά. Σας δίνω ευθύ αμέσω το λόγο κύριε Πίτροπε και συνέχεια θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή ε, Αρλίν. Καλημέρα σε όλους. Με θαρρύνουν ιδιαίτερα τόσο είπε ο κύριος Ντάιμον, τον οποίο έχω συναντήσει εδώ και πάρα, πάρα πολλές φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Μολονότι ορισμένες φορές στα πλαίσια του τραπεζικού κλάδου συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν όμως πολύ σύντομη μνήμη. Και όσον με αφορά, εγώ πάντα έλεγα και πάντα έπρατα κανένα λόγος, λέγοντας ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουμε σύντομη μνήμη, να ξεχνάμε εύκολα δηλαδή τους λόγους και τις συνέπειες της τραπεζικής κρίσης. Και όπως είπατε και εσείς, χθες είχαμε την πέμπτη επέτειο από την κατάρρευση και τη χροκοπία της Lehman Brothers. Εγώ λοιπόν δεν ξεχνάω εύκολα και πραγματικά θεωρώ ότι ε, προσπαθούμε να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ότι σίγουρα όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το έργο μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυτούμε αυτή τη στιγμή. Όπως όμως είπαμε και στο G20 της Αγίας Πετρούπολης και όπως είπαμε άλλωστε και στο ΕΚΟΦΗΝ, όπου συμμετείχα το Σάββατο με την Σάρον Bowles η οποία ήταν και αυτή παρούσα, Πραγματικά πρέπει αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αντλήσουμε τα πρώτα σημαντικά διδάγματα αυτής της οικονομικής κρίσης και ότι επιτέλους η δράση μας αναγνωρίζεται. Οι παρόντες υπουργοί και διοικητές τραπεζών αναγνώρισαν πραγματικά το έργο μας και μας ενθάρρυναν να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο προκειμένου να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε μια σχετική πάντα σταθερότητα και να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον για τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να συνεχίσουμε το έργο μας από το να κάνουμε απλώς ένα απολογισμό και να επαναπαυόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στις χώρες εκείνες οι οποίες υπολείπονται στον τομέα του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέσα της ε, χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, τα οποία έχουμε προτείνει, και νομίζω ότι οφείλουμε επίσης να καταφέρουμε να καταστήσουμε πιο ισχυρό το χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα βελτιώνεται, μόλον ότι όπως σας είπα τα πάντα είναι σχετικά το επίπεδο κεφαλαιοποίησης και μόχλευσης των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών είναι πλέον συγκρίσιμο με το επίπεδο που έχουν οι τράπεζες στις ΗΠΑ και βρισκόμαστε σήμερα πέρα από τα ελάχιστα όρια τα οποία απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες όσον αφορά τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει του 11%. Νομίζω ότι τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία είχαμε στο Βίλνιους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι καθησυχαστικά. Σας είπα ότι υπολείπονται πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε ακόμα. Ξεκινώντας από μια απόλυτη προτεραιότητα, η Τραπεζική Ένωση αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό πρόγραμμα το οποίο έχουμε και το είπα και στην Ολομέλεια την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της σημαντικότατης αυτής ψηφοφορίας που έλαβε χώρα. Και είπα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά είχαμε τρεις πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Τη ψηφοφορία για την έκθεση Μακάρθη για την κατάχρηση των αγορών, τη ψηφοφορία για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και τέλος μια πολύ σημαντική ψηφοφορία όσον αφορά την εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Πρέπει επίσης να σας ότι προκειμένου να καταφέρουμε να θεσπίσουμε την Τραπεζική Ένωση στα πλαίσια της Ευρωζώνης, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει το ενιαίο αυτό εγχειρίδιο κανόνων να ισχύει τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Επίσης θα πρέπει να καταφέρουμε να θεσπίσουμε, να, καταρπί, να καταρτήσουμε αυτό το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, πράγμα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με την δέσμη μέτρων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις υπαριθμών 4 και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο κατακαιρματισμό που είχαμε στα πλαίσια του τραπεζικού τομέα. Με την δέσμη μέτρων CRD4 καταφέραμε να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τις τράπεζες, να μειώσουμε δηλαδή τον κατακαιρματισμό τους, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε για να φέρουμε πιο κοντά το τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα στην φορολογία, τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, και, το εταιρικό δίκαιο. Όσον αφορά τώρα το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, ο Πίτερ Σάιμον το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, έχουμε και την εγγύηση των καταθέσεων. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται για το ζήτημα αυτό και ιδίω για την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών. Σίγουρα πρέπει να καταβάλουμε πολύ σημαντικέ προσπάθειε για να ολοκληρωθεί το Single Rule Book, το ενίο εγχειρίδιο κανόνων και προκειμένου αυτό να αρχίσει χάρη Τραπεζική Ένωση να χρησιμοποιείται πλήρω. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία, οι συνάδελφοι Γκίγκολτ και Τάισεν εργάστηκαν πάρα πολύ για το ζήτημα αυτό και έχουμε και ένα ψήφισμα της Ελίζα Φερέιρα το οποίο θα εξετάσει η δική σας η Επιτροπή. Επίσης την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας που είχαμε, διεξήχθη μια πολύ δύσκολη θα έλεγα συζήτηση, συζήτηση γεμάτη προκλήσεις, το οποίο είναι απόλυτα λογικό για ένα ζήτημα το οποίο είναι τόσο πολύπλοκο από νομικής και νομοθετικής πλευράς. Είδα πάντως εν, είδα πολλούς υπουργούς και πολλούς διοικητές τραπεζών και θεώρησα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με την πρόταση αυτή κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ γρήγορα το δεύτερο αυτό πυλώνα στην Τραπεζική Ένωση. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν αφενός στην νομική βάση της πρότασής μας, δηλαδή το άρθρο 114, εμείς θεωρούμε με την υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι η νομική βάση του άρθρου 114, δηλαδή της εσωτερική αγοράς, είναι η πιο χρήσιμη, η πιο αποτελεσματική και λειτουργική βάση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το δεύτερο αυτό επίπεδο, το δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Σε ένα μεταγενέστερο τώρα στάδιο, σε μια μεταγενέστερη μεταρρύθμιση της συνθήκης, όπως είπε και ο Βόλφκαν Σόιμπλε, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα. Πάντως, μπορούμε με την ισχύουσα αυτή νομική βάση να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε αν μη τι άλλο με το σύστημα αυτό, να θέσουμε δηλαδή, το δεύτερο πυλώνα. Επίσης στήθηκε και το ζήτημα της δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας αυτής, καθώς επίσης τη θέση που θα έχει εξηγήνωση των τραπεζών στα πλαίσια της πρότασης. Για όλα αυτά τα ζητήματα είμαι στη διάθεσή σα προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα δυναμικό συμβιβασμό, όπω κάναμε και με το ζήτημα τη εποπτεία. Απλώ θα πρέπει να καταλήξουμε στο τέλο σε ένα σύστημα το οποίο στην πράξη θα λειτουργεί. Ένα σύστημα το οποίο θα αντλεί τελικά όλα τα διδάγματα τα οποία είδαμε από δυναμίε τη Δέξια και άλλων τραπεζών είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συντονίσουμε την δράση των εθνικών αρχών εξυγίανσης, οι οποίες δεν ήθιστε να συντονίζονται και να συνεργάζονται. Με την επιφύλαξη λοιπόν αυτή να βρούμε μια καλώς λειτουργούσα λύση, είμαι στη διάθεσή σας για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό συνεργαζόμενος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο των Υπουργών. Πέρα από την Τραπεζική Ένωση και το ενιαίο κανόνων που πρέπει να ολοκληρώσουμε, υπάρχουν και διάφορε άλλε πρωτοβουλίε, οι οποίε απασχολούν ιδιαίτερα την Επιτροπή σα. Αναφέρθηκα για παράδειγμα στην κατάχρηση των αγορών, για την οποία η κυρία Μακάρθη ε, υπέβαλε έκθεση η οποία εγκρίθηκε. Θα ήθελα πραγματικά τα κράτη-μέλη, στα οποία στοχεύω μάλιστα να στείλω και μία επιστολή, να αρχίσουν ταχύτατα να εφαρμόζουν το κείμενο αυτό για την ε, καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των, της κατάχρησης των αγορών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια πιο δεοντολογική εσωτερική αγορά. Επίσης έχουμε το ΜΥΦΙ, την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για το οποίο συγητής είναι ο κύριος Φέρμπερ. Θέλουμε και πάλι στο πλαίσιο αυτό να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε πολλές από τις δεσμεύσεις του G20. Έχουμε επίσης το Omnibus 2, το οποίο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες. Έπειτα έχουμε τον κανονισμό για το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, με εισηγητή, εισηγήτρα την Κέι Σουίνμπουρν, όπου πιστεύω ότι στα πλαίσια της Λουθανικής Προεδρίας θα καταφέρουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε, σε έναν γενικό προσανατολισμό και έπειτα έχουμε και το πρίψα για το οποίο έχουμε μία έκθεση της ε, κυρίας Περές, δέσμη επενδυτικών προϊόντων για τους ιδιώτες επενδυτές. Έχουμε επίσης την πρόταση USITS 5 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και έχουμε έπειτα και την έκθεση Κλούτε, η οποία με ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερος όσον αφορά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε έναν απλό τραπεζικό λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση ε, να καταφέρουμε να προωθήσουμε όλε τι προτάσει αυτέ οι οποίε προστατεύουν του Ευρωπαίου πολίτε και του Ευρωπαίου κατανα... καταναλωτέ. Όσον αφορά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία για τα ανυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, για την οποία η είναι ο κύριο Σάντσε Πρεζέντο, πρέπει να πω ότι και το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Υπάρχουν βέβαια και διάφορε άλλε προτάσει που έχουν να κάνουν με τι λειτουργίε του χρηματοπιστωτικού συστήματο θα μπορούσα να αφαιρθώ πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές. Συγκρισιμότητα και διαφάνεια όσον αφορά τα τραπεζικά τέλη, η απλούστευση της κινητικότητας και της αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών, οι υπηρεσίες πληρωμών, η πλαισίωση των δικτών αναφοράς ή επίσης και μια πρόταση την οποία ξεκίνησα αρκετά πρόσφατα όσον αφορά το παράλληλο, το παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο θέλει να υποβάλει μία πρόταση Όσον αφορά τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στην έκθεση Λίκανεν για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, η έκθεση πρωτοβουλίας ε, της ε, Προέδρου σας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο. Τέλος κυρίες και κύριοι θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζεται από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η οποία συμμετέχει και αυτή με τη σειρά της το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο εποπτείας και διαφάνειας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, μεταρρύθμιση του ελεγκτικού τομέα, ενίσχυση των κανόνων όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα ήθελα επίσης να ολοκληρώσω την ομιλία μου αυτή αναφερόμενος ε, σε όλες αυτές τις ε, νομοθεσίες, σε όλες αυτές τις νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει πραγματικά να επικεντρώσουν περισσότερο τις προσπάθειές μας στο παραγωγικό κεφάλαιο και όσο τόσο στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η νέα αγορά να έχει πιο υγιείς και πιο διαφανείς πλέον βάσεις και να καταφέρουμε τελικά να ε, αναγκάσουμε, αν θέλετε, την χρηματοπιστωτική αγορά, τις χρηματοπιστωτικές αγορές να εξυπηρετούν τον Ευρωπαίο πολίτη, τους καταναλωτές και να μην επικεντρώνονται μόνο στα δικά τους συμφέροντα, όπως έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Όσον αφορά τώρα την πράσινη βίβλο για τις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ε, λάβαμε πάρα πολλές αντιδράσεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Ε, αναλύουμε τώρα τις αντιδράσεις αυτές, απαντήσεις αυτές και θέλουμε να καταλήξουμε τελικά σε κάποιες προδραστικές νομοθετικές προτάσεις, όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν με το διαβατήριο για, το, για τα επενδυτικά κεφάλαια ή αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν με το cloud founding. Θα ήθελα εν τέλει κυρίες και κύριοι να σας πω ότι ε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να επαναπαυτούμε, δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Αντίθετα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε δράση. Ξέρετε ότι ε, τα περισσότερα από τα κείμενα στα οποία αναφέρθηκα μόλις τώρα αρχίζουν και εφαρμόζονται και υλοποιούνται, πέντε χρόνια μετά την υπόθεση των Lehman Brothers και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι πλήττονται ακόμα από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό λόγο λοιπόν θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να είμαστε συνεχώς σε ετοιμότητα, να αναλαμβάνουμε δράση, γιατί Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε από πολιτική πλευρά να αντιμετωπίσουμε τι λαϊκίστικε τάσει που βλέπουμε σε πάρα πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Okay, uh, Μάλιστα. Συνάδελφοι, 17 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Θέλω να θέσουν ερωτήσεις στον Επίτροπο. Αν λοιπόν να τηρήσουμε τους κανόνες που έθεσαν οι συντονιστές, θα πρέπει έχουμε μία ώρα και 25 λεπτά, 5 λεπτά για κάθε έρωτα απάντηση. Ξεκινούμε από το ΕΛΚ και το Ζαν Πολ Σε 5 λεπτά θα πρέπει να διεκπαιρεώνουμε κάθε ερώτηση με την απάντησή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολύ σωστά είπατε ότι δεν θα πρέπει ούτε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, ούτε να κάνουμε απολογισμούς. Γιατί με τους απολογισμούς ε, χάνουμε χρόνο από το έργο που πρέπει να κάνουμε τους λίγους μήνες που μας έμειναν. Αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πόσα έχουμε κάνει ήδη. Γιατί μας υπενθυμίσατε τα διάφορα κείμενα που ξεκίνησαν ε, και πολλά διεκπαιρεώθηκαν μετά από στενή συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με φυσικά το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και έχουμε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για όσα έγιναν, αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει. Οπότε είναι λογικό να τονίζουμε τον ε, εξάρχοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει μια τάξη σε αυτή την κρίση. Και όπως είπατε κι εσείς, ε, για να ξαναφέρουμε τα πράγματα στη σωστή τους ε, τροχιά και ειδικά να απαντήσουμε σε αυτούς που λένε ότι η υπερβολική ρύθμιση σε κάποια περίπτωση είναι αυτό που επιδιώκει η Ευρώπη, γιατί το αντίθετο μας έφερε στην κρίση που είχαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που έγινε του αμερικανικού τραπεζικού τομέα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Γιατί πολλές φορές διαβάζουμε παρά όσα έχουν ε, γίνει από κάποιου παρατηρητές που υποτίθεται ότι είναι έγκυροι, ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας είναι ασθενέστερος από τον αμερικανικό. Εσείς ε, τι γνώμη έχετε για το θέμα αυτό. Θαυμάσια. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για την απάντηση. Ε, πολύ σημαντική ερώτηση θα πρέπει φυσικά να έχουμε υπόψη τις διαφορές μεταξύ του Αμερικανικού και του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και τον τρόπο που τον, τους αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας, που είναι πολύ μόρφος, χρηματοδοτεί το 75% της οικονομίας μας. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς εφαρμόζουμε τους κανόνες της Βασιλείας. Και ε, σε 8.300 τράπεζες με βάση την CRD4. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν ε, σε 30, μόνο τράπεζες του κανόνες της Βασιλείας. Εμείς σε 8.300 τράπεζες τους κανόνες της Βασιλείας και τις τέταρτες οδηγίες για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις. Τώρα υπάρχει το θέμα των συνθηκών, ε, ε, συνθηκών θεμητού ανταγωνισμού και της αμοιβαιότητας, γιατί υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των τραπεζών μας και των Αμερικανικών τραπεζών. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το νέο επόπτη που θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που έχουμε συστήσει, ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός τομέας έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Τα ίδια κεφάλαια έχουν ε, σημειώσει πρόοδο και για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες ε, το καλύτερο το πιο ποιοτικό κεφάλαιο φτάνει στο 11% και μάλιστα έχω και κάποια αριθμητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της ΕΜΠΑ, που λέει ότι εφ' εξής, σε ό,τι αφορά το πιο ποιοτικό κεφάλαιο, ε, έχουμε ξεπεράσει τα ελάχιστα 400 δισεκατομμύρια πάνω από 7% και 200 δισεκατομμύρια πάνω από 9% που είναι τα ποσοστά που ορίστηκαν πέρυσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα ποσοστά είναι 13,5% στι ΗΠΑ Πολιτείες και 2,65%. Τώρα level ratio 3,88% και 3,61 αντίστοιχα στην Ευρώπη. Τώρα, weighting assets, accounting assets, ε, ε, ratio 34-32. 34 Ηνωμένες Πολιτείες, 32 στην Ευρώπη. Αυτά λένε τα στοιχεία και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους και από την κατάσταση αυτή που είναι συγκρίσιμη θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε γιατί πέρα των μεγάλων τραπεζών έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ μικρές τράπεζες γιατί από τις 8.000 μερικές είναι πολύ μεγάλες ε, είτε εθνικές ή πολυεθνικές, είτε ατλαντικές, αλλά δεν είναι όλες πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε αυτά τα τεστ προσωμείωσης ακραίων συνθήκων και η αξιολόγηση που θα έχουν πορίσματα που θα είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Θαυμάσια καταφέραμε να τηρήσουμε το πεντάλεπτο στην πρώτη ερώτα-απάντηση. Ο Πίτερ Σάιμον, τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι ε, παρουσιάσει σα σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Μία ερώτηση να σα κάνω σε ό,τι αφορά την γερμανική τοποθέτηση. Το ερώτημα του πόσο μπορούμε να επιβαρύνουμε το φορολογούμενο, πόσο μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία καλή πρόταση για το ταμείο αυτή και το μηχανισμό αυτή ε, εναλλαγής. Έτσι θα είχαμε την ευκαιρία με ένα ενιαίο ταμείο, με ένα ενιαίο κανονισμό να μπορέσουμε να πετύχουμε και πάλι μια ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η γερμανική κυβέρνηση αντιτάσσεται. Έχει ε, τέτοιες αμφιβολίες που δεν έχει Κανένα άλλο εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δήλωσε ότι αυτές οι νομικές αμφιβολίες είναι πολιτική φύσεως. Η Γερμανία είναι μια κυβέρνηση που μπλοκάρει τον φορολογούμενο για να μπορέσει επιτέλους να ξεκινήσει μια νέα πορεία παρά τον ενιαίο αυτό δρόμο έχουν δηλώσει ότι η πρόταση αυτή θα, η πρόταση αυτή θα τύχει τη υποστήριξή σα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τι αμφιβολίε αυτέ τη Γερμανία λαμβάνετε υπόψη, μεν, αλλά θα συνεχίσετε παρά τι ενστάσει αυτέ. Ή η Γερμανία με το μπλοκάρισμα αυτό που προκαλεί θα κοστίσει, αν θέλετε, στο γερμανό φορολογούμενο και στους υπόλοιπους φορολογούμενους. Καταρχήν, Τραπεζική Ένωση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε κάθε φορά όσο βάση θα έχει το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Και παραλαμβάνω αυτό που είπε και στην εισαγωγή μου ότι πρώτα χρειαζόμαστε το κοινό εγχειρίδιο κανόνων και μετά θα μπορέσουμε να συστήσουμε την Ευρωπαϊκή, Τρα... Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Γιατί τι θα πει η Τραπεζική Ένωση. Εφαρμόζουμε στην τράπεζα τους κανόνες εποπτείας και εξυγίανσης που ισχύουν ήδη για τους 28 χώρε και θέλουμε με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό και σχεδόν ομοσπονδιακό τρόπο να τις εφαρμόζουμε στην Ευρωζώνη που εκεί υπάρχει συστημικός κίνδυνος και αλληλεξάρτηση των τραπεζών και πολύ άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ των κρατών και των τραπεζών. Ενιαίο λοιπόν χειρίδιο κανόνων είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και φυσικά εκεί έχουμε και την ε, οδηγία για την εξηγήση και το κείμενο για την εγγύηση καταθέσεων. Η Τραπεζική Ένωση έχει δύο πυλώνε. Ο πρώτο είναι η υποπτία, και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίσατε αυτή την έκθεση την περασμένη εβδομάδα και σα ευχαριστώ θερμά. Ε, ακούστηκαν κάποιες επιφυλάξεις, ε, επικρίσεις ε, και διστάμενες απόψεις στην πρότασή μου για την εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Θα θυμάστε και στην δική σας χώρα ακούστηκαν επικρίσεις και δεν ερμηνεύτηκε τελικά αυτή η πρόταση ως μπλοκάρισμα. Φυσικά θέλουμε μια ασφάλεια δικαίου και αντιλαμβάνομαι αυτό σας το μέλημα και θα είμαστε προσεκτικοί γιατί θέλουμε με τα κείμενά μας να διασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια δικαίου. Ο δεύτερος πυλώνας είναι σημαντικός και τον προτείναμε ε, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίασης των Τραπεζών. Φυσικά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αρχή αρμόδια για την εξυγίαση και τη δυνατότητα να αποφασίσουμε και κατεπηγόντως την εξυγίαση τραπεζών με αποτελεσματικό τρόπο. Οφείλω να ομολογήσω και θα σας τα πω ειλικρινά δεν εξέφρασε κάποια αντίδραση ή αντίθεση η γερμανική κυβέρνηση για το κείμενο αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και ενδιασμοί με βάση κάποια νομικά στοιχεία και φυσικά θα ζητηθεί η νομική υπηρεσία, αλλά η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ε, έδωσε θετική γνωμοδότηση για την ε, νομική βάση, το άρθρο 114 που σας ανέφερα. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε λύση. Και είπα ότι σε ένα δεύτερο, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, από τη στιγμή που θα έχουμε με βάση το 114 θεσπίσει αυτή την αρχή εξυγίασης, φυσικά θα βελτιώσουμε την ικανότητά μας για εξυγίαση. Και αν δεν θέλω να δεσμεύσω εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το μηχανισμό σταθερότητας γίνει ένα κοινοτικό όργανο, κοινοτικό μηχανισμός, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, αργότερα μπορεί και αυτός ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας να έχει την ικανότητα εξυγίασης. Αλλά αυτή τη στιγμή υπόκειται στην διακυβερνητική ε, λειτουργία και χρειάζεται ομοφωνία. Στο Blueprint πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Ευρωζώνη και με την αλλαγή των συνθήκων τροποποιούμε το νομικό αν τροποποιήσουμε το νομικό καθεστώς του μηχανισμού σταθερότητας θα μπορέσουμε να το τροποποιήσουμε και να περιλάβουμε και την εξυγίαση στο έργο του. Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε αλλαγή των συνθήκων για να λειτουργήσουν όλα αυτά γιατί ε, δεν θέλουμε να επαναληφθεί η τράπεζα και στόχος της εξυγίασης είναι οι τράπεζες να αναλαμβάνουν το κόστος ε, των λαθών τους και όχι οι φορολογούμενοι. Επίσης, ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις κυβερνήσεις. Άλλωστε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την άποψη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Να δώσουμε λίγο παραπάνω, ε, παραπάνω δευτερόλεπτα σε εσά λόγω της ημέρες. Ο κύριος Κλίνης από πλευρά τη Άλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Να μείνουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Το θέμα δεν είναι αν χρειάζεται νέα συνθήκη ή όχι. Το θέμα είναι το εξή. Το Ταμείο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Δεν έχει ακόμα ε, λάβει, ας πούμε, κονδύλια. Θα πάρουν πολλά χρόνια αυτά. 50 έως 60 δισεκατομμύρια χρειαζόμαστε προκειμένου να έχουμε δυνατότητα ε, για μια μεγάλη τράπεζα. Προτάθηκε το Σάββατο από το Ράσμουσεν να υπάρχει ο μηχανισμός σταθερότητας, το ESM, να χρηματοδοτήσει αυτό το κενό. Τι πιστεύετε για την πρόταση αυτή, κατά δεύτερον. Δεν είναι θέμα μόνο χρηματοοικονομικό, το θέμα είναι και η θέληση που υπάρχει να βοηθήσουμε χρηματοπιστωτικά τέτοια ιδρύματα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα ιδρύματα, αλλά η FDIC παράλληλα δεκάδες τέτοια ιδρύματα έχει βοηθήσει. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε να γίνεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Υπάρχει βούληση για να δώσουμε για παράδειγμα ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Και κατά τρίτον, διαπιστώνω ότι όλο και πιο πολλές δραστηριότητες από τον κλασικό ε, ε, τομέα χρηματοπιστωτικών έχουν περνάνε στον σκιώδη, αν θέλετε, κλάδο σε ό,τι αφορά τα ε, παράγωγα, για παράδειγμα, που είναι πάνω από 50% και έχουν περάσει στον πιο σκιώδη κλάδο. Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα? Ε, ε, Κύριε Κλίντς, προφανώς απαιτείται χρόνος για να βρεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Αν όμως δεν δημιουργήσουμε το Ταμείο αυτό, τότε θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε το ακόλουθο. Αν θεωρούμε ότι η ιδέα αυτή είναι σωστή, να δημιουργήσουμε δηλαδή το ταμείο αυτό για να καταφέρουμε τελικά διασνοριακά να εξηγιαίνουμε τις τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνεται αυτό μέσω ενό ταμείου, εμένα αυτή είναι η απόψή μου και νομίζω ότι δεν, κανείς, δεν μπορεί κανεί να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή προτείνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρόταση αυτή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα δέκα χρόνια και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια σωστή λειτουργία του, τομή, του Ταμείου αυτού. Πρόκειται για ιδιωτικού πόρου που θα χρηματοδοτήσουν το Ταμείο αυτό. Στο ενδιάμεσο ε, διάστημα πρότεινα και εγώ ότι θα μπορούσαμε όντως να δανειστούμε κάποιους πόρους και να τους αποπληρώσουμε στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους. Θα μπορούσαμε πάντως να φανταστούμε και αυτό το ενδεχόμενο, να δανειστεί το ταμείο αυτό από τις αγορές για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του εφόσον αυτό κρυθεί αναγκαίο. Δεύτερον, ναι όντως, θεωρώ ότι με την οδηγία για την εξυγίανση τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εξηγαίνουν ε, το τραπεζικό τους κλάδο. Και με την Τραπεζική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα γίνεται με έναν τρόπο συλλογικό και αποτελεσματικό. Αντί να κινούμαστε ο καθένας κατακαιρματισμένα, μεμονωμένα, σε έκτακτες πλέον περιπτώσεις και χωρίς να υπάρχει καμία ευελιξία. Νομίζω λοιπόν ότι με την οδηγία αυτή για την εξυγίανση από τη στιγμή που θα αρχίσει να εφαρμόζεται θα και με τη βοήθεια του Ταμείου θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρούμε σε μια σωστή, σωστά διαρθρωμένη εξυγίανση, σε μια τακτική εξυγίανση. Ξέρετε ότι κοστίζει πολύ λιγότερο να προλαμβαίνει κανείς τις δυσάρες καταστάσεις, είναι πολύ σημαντικότερο να επενδύει κανείς στην πρόληψη από το να πρέπει στη συνέχεια να διορθώνει τα κακό κείμενα. Αυτό το έχουμε δει σε όλη αυτή την περίοδο των τελευταίων πέντε ετών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την εξυγίανση αυτή των τραπεζών. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα εκ των προτέρων. Θα μπορούσα να μιλήσω και για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και εγώ ανησυχώ για τα φαινόμενα στα οποία αναφερθήκατε. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν την ρύθμιση του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε να ασχολούμεθα με την ρύθμιση των πόρων αυτών που κινούνται στον παράλληλο τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε οι οποίοι όντω ενδεχομένω να κινηθούν προ τον κλάδο αυτό για να αποφύγουν τον πλέον ρυθμισμένο κλασικό τραπεζικό τομέα. Um, uh, Μετά έχουμε τον κύριο από το ECR. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επιτροπό. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την κατάρρευση της Lehman Brothers 15 Σεπτεμβρίου του... και υπάρχουν τρεις αρχές που... Τρία θέματα που δεν έχουμε κοιτάξει. Καταρχάς δεν βλέπουμε, δεν θέλουμε να σταματήσει η εξυγίανση, τη διάσωση των τραπεζών από του προλογούμενου, κατά δεύτερον θέματα ευθύνη και τρίτον σε ό,τι αφορά τα λογιστικά πρότυπα. Τι γίνεται. Μιλάτε για τι υπηρεσίε τις υπηρεσίες και πώς επιβαρύνονται σε ό,τι αφορά την τραπεζική ε, μεταρρύθμιση. Πραγματικά όμως αυτό πρέπει να γίνει και το ξέρω ότι σας έχουν ασκήσει λόμπι οι τράπεζες, αλλά είμαι βέβαιος ότι και οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου όταν σα παρατηρούν να προχωρήσετε με το θέμα αυτό. Και θα ήθελα λοιπόν να σα Δεν θα σα ρωτήσω για την καθυστέρηση. Να έρθω όμω στο τρίτο θέμα. Οι ανησυχίε πολλών επενδυτών για τα λογιστικά πρότυπα IFRS. Ξέρετε και ξέρω κι εγώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η σχετική επιτροπή, η Τράπεζα τη Αγγλίας και μεγάλε τράπεζε θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα με το IFRS. Εδώ στο Κοινοβούλιο σε μία σειρά εκθέσεων έχουμε εκφράσει συνένεση ε, από όλο το πολιτικό φάσμα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι θα ήθελα να ρωτήσω αν ο Επίτροπος ε, θα εξετάσει την άλλη ανησυχία του κατά πόσο το IFRS συνάδει με το εταιρικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι Υπάρχει μια σχετική γνωμοτότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη συμβατότητα αυτή, τη μη συμβατότητα αυτό. Και επίση για, τα... για την τάση σύγκληση σε ό,τι αφορά τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορούν πιο πολύ την ενημέρωση με τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με, την... Ε, με κανόνες που υπάρχουν και τα πώ ακολουθούνται. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ε, ε, Κύριε Καμάλ. Μίλησατε για τρεις αρχές. Αν το κρίνετε χρήσιμο θα το επαναλάβω. Ακούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, τραπεζίτες ε, και άλλους και δεν πρόκειται να υποκύψω σε κανένα λόμπινγκ, σε καμία ομάδα πίεση, σε καμία πίεση. Και χαίρομαι που με την ε, συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα είναι πιο ισορροπημένη ε, και θα έχουμε και τη Finance Watch που θα μπορεί ίσως να μας δώσει μια ανεξάρτητη γνώμη για τη, την νομοθεσία που ετοιμάζουμε και να μην έχουμε μόνο την γνώμη των τραπεζών. Οι τρεις αρχές θα εφαρμοστούν. Αυτούς, αυτές θέλουμε να εφαρμόσουμε, να προστατεύσουμε τον φορολογούμενο. Το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία ε, και στην προηγούμενη ε, απάντηση προς τον κύριο Κλίντς. Έχουμε πια τους μηχανισμούς εφόσον ψηφιστούν για να εξηγαίνουμε τράπεζες χωρίς ε, να χρειαζόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων. Και αν όλα τα κείμενα που σχεδόν όλα έχουν ε, ψηφιστεί, αν λειτουργούσαν ήδη, αν είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, κάνοντας μια προσωμείωση, ε, με διαφορά 34 εξαιρέσεων, όλες οι περιπτώσεις τραπεζικής κρίσης όπου χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα φορολογουμένων τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν θα ήταν αναγκαία θα είχαμε τις κρίσεις, αλλά θα τις αντιμετωπίζαμε διαφορετικά και όχι με χρήματα των φορολογουμένων, με τρεις-τέσσερις διαφορές, τις τρεις-τέσσερις εξαιρέσεις. Και βλέπετε πόσο θα ε, βελτιωθεί η κατάσταση εφόσον ε, αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα κείμενα. Σε ό,τι αφορά τι ευθύνε, ε, αυτό κάνουμε και με την οδηγία για την κατάχρηση των αγορών, χειραγώγηση αγορών. Και θα επεκταθεί αυτή η ευθύνη και μάλιστα μεθαύριο θα υποβάλω το κείμενο εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκριτικό κανόνα, το benchmark. Και όσοι έκαναν κάποιε καταχρήσει του benchmark θα υπάγονται στην οδηγία και για την κατάχρηση των αγορών και στο επόμενο κείμενο για τι ποινικέ κυρώσει του στέλνουμε και φυλακή. Οπότε θα έχουμε μια διεύρυνση τη ευθύνη. Το ίδιο έγινε και για τους ε, οίκους ε, αξιολόγησης. Με τη δημιουργία benchmark θα πρέπει να δούμε και ποιοι ε, μηχανισμοί δημιουργούν αυτά τα benchmark, του συγκριτικού κανόνε. Δεν του κατηγορούμε, αλλά θέλουμε να υπάγονται και αυτοί στη μεθοδολογία, στη διαφάνεια και στην εγκυρότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούν. Θα πρέπει και αυτοί να φέρουν τι ευθύνε του. Ένα άλλο σημείο για τους λογιστικούς κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα. Για τους γνωστούς λόγους πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναθέσει αυτό το θέμα σε ένα διεθνή οργανισμό που ονομάζεται EASB και έχει έδρα στο Λονδίνο. Εγώ από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Επίτροπος συμμετείχα τακτικά στις συνεδριάσεις της EASB, αυτού του φορέα και αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο θέμα της διακυβέρνησης και την ανάγκη της βελτίωσης γιατί είναι ένα World of trust της EASB, μια τεχνική ομάδα και ευτυχώς τελικά συστήσαμε και ένα συμβούλιο εποπτείας κατά κάποιο τρόπο παρακολούθησης που εκπροσωπούνται και τα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Πάντως εγώ είμαι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το, ESB, σε αυτό το φορέα. Βελτιώθηκε λοιπόν ο διάλογος μεταξύ του ESB και του Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου Μιλήσαμε πολύ για τη διακυβέρνηση και την ανάγκη βελτίωσή τη. Τώρα θα πρέπει να εγγύψουμε στη ποιότητα των λογιστικών κανόνων. Και εκεί υπάρχει η κλασική αντιπαράθεση μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων σε ό,τι αφορά τη θέση που θα δώσουμε στην, ε, στο market value ή στη σωστή αξία. Η τιμή της αγοράς δεν είναι ίδια με την ε, σωστή τιμή, τη δική τιμή θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και εγκυρότητα στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Αν εφαρμόσουμε στην αρχή της σωστής τιμής ε, ε, απερίσκεπτα, όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί μερικές φορές, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα των αγορών ε, και αβεβαιότητα στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επιδιώκουμε μια μεγαλύτερη σύγκληση και δημιουργήσαμε τα πρότυπα EFRS, που είναι τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικών αναφορών. Είναι μια συμβεστική λύση που όμως δεν εφαρμόζεται με του Αμερικανού. Και είπα πρόσφατα στο Δικαιτικό Συμβούλιο του ISB ότι η ευρωπαϊκή υπομονή έχει και τα όρια της και ότι τα όρια αυτά σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Αυτή είναι και η γνώμη μου. Και θα ήταν κρίμα οι εταίροι τη, τη να επανέλθουν ε, στα θέματα της κυριαρχίας ό,τι αφορά τους λογιστικούς κανόνες γιατί στόχος των δίκαιων συναλλαγών ε, παγκοσμίω είναι η σύγκληση και γι' αυτό συστήσαμε και την νέα για τη σύγκληση. Κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή και ελπίζω με την, με τη νέα πρόεδρο της CFTC, της ISCC με την οποία μα, ε, είχα συζητήσει, ελπίζω λοιπόν η νέα πρόεδρος ε, να αλλάξει θέση. Ο κύριος Λάμπερτς από τους Πράσινους. Κύριε Πίτροπε, καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε και όντως βλέπουμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Πρώτη παρατήρηση είπατε ότι θα αρχίσουμε να εφαρμόσουμε τη Βασιλεία Παριθμών 3 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγώ θα σας πρότεινα να προτείνετε την ε, εφαρμογή της Βασιλείας 3 ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά αυτόν τον τρόπο ενδεχομένω να καταφέρουμε να αποκομίσουμε περισσότερα έσοδα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αστευόμενος τα όλα αυτά. Είπατε επίσης ότι ε, πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να αυξήσουμε το επίπεδο και το πετύχαμε αυτό ε, των κεφαλαϊκών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρ' αυτά υπάρχουν ακόμα κάποιοι κίνδυνοι. Οι ε, μεγάλες συστημικές τράπεζες ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή παίζουν πάρα πολύ με τη στάθμιση του κινδύνου. Και πολύ συχνά όταν ξύνουμε λίγο την επιφάνεια βλέπουμε ότι ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιε βελτιώσει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, από την άλλη όμως να έχουν γίνει απαραίτητε διορθώσεις όσον αφορά τη στάθμιση των κινδύνων. Και δεύτερον, πολύ συχνά βλέπουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένε ευρωπαϊκέ τράπεζε οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα πολύ σημαντικά προβλήματα και να μην ανταποκριθούν στο λεγόμενο quality review, σε αυτήν την αναθεώρηση ποιότητας την οποία πρέπει να κάνουμε. Αν κάνουμε αυτή την ε, αξιολόγηση ποιότητα, ενδεχομένω να καλύψουμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ θετικά και ότι τελικά τα χρήματα τα οποία έχουμε στο διαθέσιμο ταμείο, το μελλοντικό, δεν θα αρκούν για να εξηγιάνουμε τι τράπεζε. Θα καταφέρουμε να δούμε τελικά ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο δεν θα έχουμε καμία λύση δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένω να πληγεί ακόμα και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τομέα, μολονότι έχουν γίνει κάποια stress test τα οποία έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα πραγματικά να μα πείτε τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίσει με ολοκληρωμένο τρόπο να εποπτεύει με λαθασμένο τρόπο τι τράπεζε, τότε νομίζω ότι η αξιοπιστία του όλου συστήματο τίθεται ένα αμφιβόλο. Επίτροπος. Κοιτάξτε, περιγράψτε τα πράγματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο δεύτερο τμήμα της ερώτησής, της, ερωτη, της ερώτησής σας και όντως ήσασταν σωστό στον τρόπο που α, τοποθετηθήκατε. Τώρα όσον αφορά το πρώτο σας σχόλιο δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπατε για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο καθένας καλεί την επιτελέσει το έργο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σημαντικό όσον αφορά τους Αμερικάνους είναι να έχουμε μαζί τους ένα συγκρίσιμο συντονισμένο σύστημα ένα σύστημα αντίστοιχο και ένα σύστημα διαλειτουργικό αυτή την ε, διαλειτουργικότητα στο ρυθμιστικό μας σύστημα, το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις αγορές στην διεθνή αυτή εμπορική συμφωνία την οποία τώρα διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση αμοιβαίω στις αγορές μας αν δεν έχουμε αντίστοιχα διαλειτουργικά τραπεζικά συστήματα όσον αφορά συγκεκριμένα τη ρύθμιση των τραπεζών. Μπορούμε επίσης να αναφερθούμε περισσότερο και στα προβλήματα που έχουμε με τις αμερικανικές εκείνες τράπεζες που δεν είναι στην πραγματικότητα αμερικανικές, απλώς βρίσκονται σε αμερικανική επικράτεια. Πάντως μπορούμε όντως να αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό το οποίο θίξετε, δηλαδή το πόσο πραγματικά ισχυρές είναι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές τράπεζες και εμένα με απασχολεί το ζήτημα αυτό και γι' αυτό το λόγο είπα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το νέο ρόλο που θα αναλάβει στα πλαίσια του ενιαίου ποπτικού μηχανισμού για τον οποίο προετοιμάζεται πάρα πολύ σοβαρά και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Ντράγκελα και τον Προεδρεύοντα της Λιθουανικής Προεδρίας στα πλαίσια λοιπόν αυτού του νέου μηχανισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση, να έχουμε μια ακριβή απογραφή της ε, κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των κεφαλαίων των τραπεζών και να δούμε επίσης ε, πώς διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους αυτά, τα περιουσιακά του στοιχεία. Και νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πραγματικά πρόκειται με απόλυτη αυστηρότητα και σοβαρότητα να επιτελέσει το έργο της αυτό και θα καταφέρει παράλληλα να αναλύσει και τους κινδύνους οι οποίοι υφίστανται όσον αφορά τους ιδίους πόρους. Το ερώτημα το οποίο θέσατε πολύ σωστά είναι σαφώς τι θα γίνει αφού κάνουμε την απογραφή αυτή. Και τους υπουργούς τους απασχολεί το ερώτημα αυτό. Δηλαδή το ότι θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτό το οποίο ονομάζουμε backstop, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις τράπεζες όταν παρουσιαστούν ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Γιατί όταν θα γίνει αυτή η ποιοτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, προφανώς θα εντοπίσουμε και κάποιες τράπεζες με αδυναμίες. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ από το EFD. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε Μπαρνιέ. Ένα προβληματικό στοιχείο στην Τραπεζική Ένωση είναι το θέμα του κατά πόσον ε, οι ε, χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση χειρότερα θα έχουν το περιθώριο προκειμένου να κάνουν ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν ξέρουν πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη σε κεφάλαιο. Είναι πραγματικά βασικό να μας πούν και να γίνει σωστή κατανομή του λογαριασμού την εξή ερώτηση να σας κάνω. Τι δυνατότητες υπάρχουν για τις, ε, τα πολιτικά μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προκειμένου πριν να γίνει η Τραπεζική Ένωση, να έχουμε μια ρεαλιστική αξιολόγηση του κόστους και του κεφαλαίου που χρειάζεται και επίσης ό,τι αφορά τη δημοσίευση μια σχετική δημοσίευση του θέματο αυτό για έναν μηχανισμό early intervention, ε, έγκαιρη προειδοποίηση και παρέμβαση. Ε, πώς ε, αξιολογείται αυτό το θέμα. Ή πιστεύετε ότι ο λογαριασμό θα έρθει στο τέλο, όταν θα έχουν μπει οι τράπεζε στην Τραπεζική Ένωση όπου και φυσικά θα είναι πολύ άσχημη η κατάληξη. Να μου πείτε ποια είναι η απάντησή σα σε αυτά, παρακαλώ. Κύριε Μπέλτερ. Το θέμα είναι ότι στη συζήτηση αυτή θα θέλαμε όλα να γίνουν αμέσως και να λειτουργήσουν εύρυθμα και πλήρως. Βέβαια, ο χρόνος της δημοκρατίας ε, είναι πιο αργός από το χρόνο της αγοράς. Χρειάζεται χρόνος για να ψηφιστεί το κείμενο, για να τεθεί σε εφαρμογή, ε, τα τεχνικά μέσα είναι μια διαδικασία να το γίγνεστε, παρόλο που βαίνουμε με μεγάλη ταχύτητα, όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Γκοζές. Αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να πρικοδοτήσουμε με 50-60 δις ε, το Ταμείο Εξυγίασης. ή να ε, είναι σε καλή κατάσταση όλες οι τράπεζες. Θα χρειαστεί χρόνος και γι' αυτό. Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Το ενιαίο χειρίδιο κανόνων και το νομοθετικό κείμενο για την εγγύηση καταθέσεων και την εξηγήση γιατί η Τραπεζική Ένωση είναι εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα. Στα, στα πλαίσια της εποπτείας του πρώτου πυλώνα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σταθερές ε, και αυστηρές βάσεις ε, θα ξεκινήσει την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείου του ενεργητικού, φυσικά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή των Τραπεζών, που θα κάνει τα τεστ ε, προσωμείωσης ακραίων συνθήκων στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενίας αγοράς. Δεν μ' αρέσουν οι ούτε θα ήθελα να κάνω προβλέψεις για τις ανάγκες που θα έχουν οι τράπεζες της Ευρωζώνης για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Φυσικά θα χρειαστούν κάποια κονδύλια, αλλά ας μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ε, με το τομείο Ανακεφαλαιοποίησης ε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, ακόμη και πριν την Βασιλεία Φυσικά χρειάστηκαν μερικέ εκατοντάδε δισεκατομμύρια που τελικά βρήκαν οι τράπεζε με δική του αναδιάρθρωση από τι αγορέ. Τα κατάφεραν. Α μην πιθανολογούμε τώρα για τα ποσά, αλλά αν χρειαστούν ανασταλτικοί μηχανισμοί backstop σε ορισμένε περιπτώσει, το το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να προβλέψουμε τέτοιου ανασταλτικού μηχανισμού ε, δημόσιου ε, όπου χρειαστεί. Αυτά στα πλαίσια μια γενική στρατηγική. Αλλά θα δούμε τα πράγματα το καθένα στον καιρό του. Μπορεί να μην σας αρκεί τελικά αυτή η απάντηση κύριε Μπέλντερ, αλλά αυτό που κάνουμε δύσκολο είναι και χρονοβόρο. Θα προσπαθήσουμε με νυφαλιότητα και διάβια να βρούμε τα πράγματα, αλλά σίγουρα η τωρινή κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί εκεί κάθε χώρα ήταν αφημένη στη μοίρα της ε, μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια θέματα και οι τράπεζες που είχαν δυσκολίες, ε, δημιουργούσαν δυσκολίες και στις υπόλοιπες, ενώ τώρα δημιουργούμε θεμέλια, ουσιαστικά επανάσταση για την Ευρωζώνη. Η Τραπεζική Ένωση είναι επανάσταση και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το να αφήνουμε το καθένα στη μοίρα του, όπως το είδαμε και με τις συστημικούς κινδύνους και συνέπειες είχε μια τέτοια κατάσταση ο κ. Μάρτιν από για Όσο ε, είμαι εδώ πέρα στο κοινοβούλιο, όσο πιο πολύ είμαι εδώ πέρα στο κοινοβούλιο, τόσο πιο πολύ με ανησυχεί η επιρροή των ε, λόμπι στη λήψη αποφάσεων. Έχουμε 700 λόμπι εδώ στους Βρυξέλλε για χρηματοπιστωτικό κλάδων με 300 εκατομμύρια ε, προπολογισμό το χρόνο. Το γνωρίζουμε αυτό. Επίση, ξέρουμε ότι πολλέ πιέσει δέχεται από λόμπι η Επιτροπή, ιδιαίτερα στο δικό σα κλάδο. Μπορείτε να μα πείτε κατά πόσον θα μα. Ε, είσαστε υπέρ της καταχώρησης όλων των επαφών με τα λόμπι και σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους για το πόσο τους μιλάτε, γιατί τους μιλάτε, πότε συναντιέστε και επίσης, ε, δεύτερο θέμα, θα δημοσιεύσετε τις παρεμβάσεις και την επιρροή των λόμπιν στις νομοθετικές ε, προτάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διατύπωση. Πολλοί συνάδελφοι προφανώς ε, θέλουν αυτό να γίνει στο Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο και στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι κάποιοι από εμάς το κάνουν αυτοθρεντικά εδώ στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου, αλλά ο Επίτροπος θα απαντήσει. Ναι, ναι, ναι, αυτό είπα λέει ο κύριος Μάρτιν. Euh, πριν από λίγο και πριν από την ερώτησή σας κύριε Μάρτιν είχα πει ότι πραγματικά έχω ακούω τους πάντες αλλά ότι δεν επηρεάζομαι εύκολα από τους λομπίστες, από τις ομάδες πίεσης. Πολλές φορές μάλιστα θεωρώ ότι είναι και κάπως αντιπαραγωγική στο έργο τους και το είπα και δημοσίως αυτό. Ε, για παράδειγμα σε σχέση με την εκστρατεία της Mastercard εξατή, ε, κατά της δικής μου της πρότασης ε, όσον αφορά τις διατραπεζικές ε, προμήθειες και τα διατραπεζικά τέλη. Ξέρετε ότι είχαν κάνει μια τεράστια εκστρατεία, είχαν πληρώσει ακόμα και ψευδή άρθρα στον τύπο, χρησιμοποίησαν ακόμα και τη φωτογραφία μου. Είδα πραγματικά τη φωτογραφία μου σε κάτι άρθρα τα οποία πλήρωνε, χρηματοδοτούσε αστικά η Mastercard και τα οποία βαίνανε κατά της δικής μου της πρότασης. Νομίζω ότι υπάρχουν και πιο ευφυείς καμπάνιες από αυτήν. Πάντως δεν επηρεάζομαι εύκολα, ούτε εντυπωσιάζομαι εύκολα. Για να είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου, με όλες αυτές τις ομάδες, κυρίως με τις ομοσπονδίες βέβαια. Κυρίως συναντιέμαι με ομοσπονδίες ασφαλιστικών οργανισμών, με ομοσπονδίες τραπεζών, γίνεται εκτενής διαβούλευση μαζί τους και μάλιστα δημοσιοποιούμε και τις γνωμοδοτήσεις τις οποίες μας υποβάλλουν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αυτών. Μπορείτε και εσείς να τις διαβάσετε στο διαδίκτυο. Δημοσιοποιούμε εκτενέστατα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία Ίσως ο κύριος Εύκοβιτς θα μπορούσε να σας απαντήσει περισσότερο για το ζήτημα της διαφάνειας. Εγώ πάντως κινούμαι δημοσίως. Το πρόγραμμά μου είναι δημόσιο, όλοι το γνωρίζουν, ε, είναι ανοιχτό προς όλους, όλοι γνωρίζουν ποιου συναντώ. Ξέρετε ότι ε, δεν προέρχομαι από τον τραπεζικό τομέα, ενδεχομένω και αυτόν είναι θετικό. Επομένως είμαι απόλυτα ανοιχτό, διαλλακτικός και αντικειμενικός αμερόληπτος όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Δεν εντυπωσιάζομαι λοιπόν, ούτε επηρεάζομαι ούτε εγώ, ούτε οι συνεργάτε μου, ούτε το γραφείο μου. Και πρέπει να σα πω και κάτι ακόμα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Πολύ συχνά, κύριε Μάρτιν, οι τράπεζε όταν υπερασπίζονται τα συμφέροντά του, ενδεχομένω να υποβάλλουν και κάποια ερωτήματα τα οποία είναι χρήσιμα και σωστά όπως για παράδειγμα κάνουν οι καταναλωτές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι μέσω της διαδικασία αυτής μας διαφωτίζουν οι ίδιοι οι λομπίστες για ένα ζήτημα. Έρχονται και μας λένε, κοιτάξτε, υποβάλλουν μια ερώτηση και εμείς λέμε, α, υπήρχε εδώ ένα πρόβλημα και δεν το είχαμε εντοπίσει. Όταν οι τράπεζες, για παράδειγμα, μας λένε ότι ε, υπάρχουν διαφορές ανταγωνιστικότητας ή ότι υπάρχει αθέμητη ανταγωνιστικότητα στις ΗΠΑ, αν οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, αρχίζουν και χρησιμοποιούν το Foreign Banking Organizations, αυτούς τους οργανισμούς, ξένους οργανισμούς ε, τραπεζών, τους ξένους τραπεζικούς οργανισμούς, τότε καταφέρνουμε και εμείς να εντοπίσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε. Εν γέννη πάντως, Πρέπει να σας πω ότι όσο δίστανται οι απόψεις, τόσο το καλύτερο στη τελευταία ανάλυση. Είναι πολύ καλύτερο να καταφέρνουμε να βελτιώνουμε τα πράγματα μέσω της αντιπαράθεσης των απόψεων. Και γι' αυτό το λόγο προωθούμε την ανταλλαγή απόψεων με όλους, αλλά και με όλους αυτούς τους ακαδημαϊκούς και τους οργανισμούς που ανεξάρτητα μπορούν να συμβάλλουν. Επερώτηση. Δεν ήθελα να αμφισβητήσω την ε, ε, ακαιρεότητά σας, γιατί είμαι πραγματικά πεπισμένος ε, από τον ρόλο σας και την ηγεσία σας στους, ε, σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους σας. Και είμαι βέβαιος και ότι η Επιτροπή θα ακολουθήσει αυτή την οδό για την αποτύπωμα των λόμπι. Μάλιστα, κυρία Βόρτμαν Κόουλ για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Είπατε και αναφέρατε πολύ σωστά τα επιτεύγματα για τα οποία έχουμε όλοι εργαστεί σκληρά σε ό,τι αφορά την πιο βιώσιμη χρηματοπιστωτική αγορά και για την εποπτεία στην Ευρώπη. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαίνεται αμφισβητεί ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας αυτής, συγκεκριμένα το να είναι ε, κάποια μέτρα κατεπήγοντα της ΕΣΜΑ για το short selling. Σε περίπτωση που το δικαστήριο λοιπόν ακολουθήσει αυτή την οδό και ο εισαγγελέα ακολουθήσει αυτή την οδό, τι θα κάνετε, γιατί τι ζητά ο εισαγγελέα η απόφαση αυτή να λαμβάνεται βάσει ομοφωνίας. Μιλάμε για κατεπήγουσες ε, καταστάσεις, κατεπήγοντα μέτρα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ε, ομοφωνία. Θα υποβάλλεται εναλλακτική νομοθεσία για να πληρωθεί αυτό το κενό στο short Ό,τι αφορά τις ανοιχτές πωλήσει η συνάδελφος, ο συνάδελφος ε, Κλίντς ε, σας ρώτησε ποιες είναι οι απόψεις σας για τις δηλώσεις Άσμουσεν πριν από κάποιες ημέρες ε, για το κατά πόσον το Ταμείο Κατεπήγοντων Μέσων μπορεί να δανείσει σε αυτό το νέο Ταμείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Κλίν, στην οποία παραπέμψατε, δεν είχαμε προτείνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι θυμάμαι, στο κείμενο που υπέβαλα για την εξυγίαση, είπα ότι στην ενδιάμεση περίοδο, όσο δεν έχει αρκετή πρικοδότηση το Ταμείο Εξυγίασης, γιατί σταδιακά θα, προσθεθεί, θα προσθεθούν κονδύλια, θα μπορούσε κανείς να δανειστεί ή να προσφύγει στην αγορά. Τώρα, αν δανειστεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα ή από ένα ευρωπαϊκό άλλο μηχανισμό, είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Και ο μηχανισμό αυτό έχει τι δικέ του μεθοδολογίες ε, ε, και θα κρίνει κατά πόσο ε, έχει νόημα να δανείσει. Είναι θέμα αμοιβαίου συμφέροντος. Πάντως σκέφτηκα ότι η ιδέα του κυρίου Άουσμουσεν θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι η μοναδική ιδέα, ίσως για να πρικοδοτήσουμε το Ταμείο Εξυγίασης με τα κονδύλια που θα χρειαστεί στην μεταβατική περίοδο, στην ενδιάμεση περίοδο. Πάντω η πρότασή του ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά όχι η μόνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα, κυρία Βόρτμαν Κόλ, αντιλαμβάνομαι και είναι και λογικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Φυσικά η νομολογία του 10 και η απόφαση, η δικαστική απόφαση έχει νομική αξία και φυσικά θα ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάσαμε προσοχή, όπως και το νομικό μου επιτελείο, τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα για τον κανονισμό Σβάρτσελινγκ ε, short selling, συγγνώμη, για τι ανοιχτέ πωλήσει που αναφέρεται το άρθρο 114 μπορεί να είναι νομική βάση για τη θέσπιση ενός οργανισμού. Και η νομολογία Μερώνη, που δεν χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μεταξύ μα, θα πρέπει να τηρηθεί πλήρωση ε, εκφέρονται ε, αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ανάθεση σε μία μόνο αρχή αυτής της αρμοδιότητας για τις ανοιχτές πωλήσει το short selling. Πάντω ε, η νομική μου υπηρεσία εξετάζει με προσοχή τα συμπεράσματα του, δικαστικού, του Γενικού Εισαγγελέα. Εμεί έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Πάντω ε, η αρχή προβλέπει ότι η δυνατότητα ε, αντίδρασης του οργανισμού είναι ο βασικός μας στόχος. Και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων ανοιχτών πωλήσεων, short selling, ο πρωταρχικός μας στόχος και θα περιμένουμε για αυτή τη δικαστική απόφαση, είναι η, δυνατότητα του οργανισμού να αναλάβει δράση εκτάκτου ανάγκη όταν υπάρχει μια κατεπίγουσα περίσταση. Τώρα δεν πρόκειται εγώ να, σχολιάσω τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέως. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, βέβαια Φυσικά δεν είναι ρόλο σα ε, να σχολιάσετε τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι αυτονόητο αυτό. Σε περίπτωση όμω που το δικαστήριο δικαιώσει τον Γενικό Εισαγγελέα, είστε έτοιμο το συντομότερο δυνατό να υποβάλλετε νομοθετική πρόταση για να καλύψετε το κενό που δημιουργείται. Γιατί είναι σημαντικό να έχει η ΕΣΜΑ αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών αυτές τις δυνατότητες δράση κατεπηγόντω ή εκτάκτου ανάγκη υπό την επιφύλαξη φυσικά τη οριστική δικαστική απόφαση. Η απάντηση είναι ναι, φυσικά θα δράσουμε αμέσω. χρειαστεί να διορθωθεί, να καλύψουμε κάποιο κενό, θα υποβάλουμε νέα νομοθετική πρόταση, φυσικά. Mr. Ο από το Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτον, τον κίνδυνο για τις δύο κουλτούρες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς ε, η Ευρωζώνη και η εκτός Ευρωζώνης και ο κίνδυνος κατακαιρματισμού. Πώς εκτιμάτε τον κίνδυνο να υπάρχει μεγαλύτερος ε, ηθικός κίνδυνο, ότι κάποιοι δηλαδή θα κρίνουν ότι κάποιο άλλο θα αποφασίσει και κάποιο άλλο θα λάβει τι αποφάσει ενώ δεν υπάρχει επαρκή επαρκής ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί, για την εξυγίανση που πρέπει να ε, γίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί τον κίνδυνο που ενέχεται να δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα παρά να επιλύσουμε άλλα ήδη υφίστανται. Δεν κατάλαβα καλά το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας. Όχι επειδή μιλήσατε αγγλικά, αλλά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους κινδύνους από ό,τι να τους αντιμετωπίσει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενδεχομένως να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις προς αυτό για να καταλάβω τελικά πού έγκυται το ερώτημά σας και ουσιαστικά ποιος είναι ο νέος κίνδυνος που ενδεχομένως εμείς να δημιουργήσουμε. Δεν εννοώ ασφαλώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει επιπλέον ε, κινδύνους. Μου αρέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνετε καλή δουλειά. Αυτό που λέω είναι ότι όταν υπάρχει νομοθεσία όταν δημιουργείται νομοθεσία που θέτει την ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξυγίανση, αλλά δεν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για την εξυγίανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε, τότε δημιουργείται ένα κίνδυνο. Όσοι τελικά αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο σε επίπεδο κράτου μέλου, ελπίζουν ότι κάποιο άλλο θα αναλάβει την ευθύνη επιλύση του προβλήματο. Και αυτό είναι μία, ξέρετε, από τι κακέ συνήθειε του ανθρώπου. Πάντα ελπίζουμε κάποιο άλλο θα αναλάβει την ευθύνη και θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Άρα αυτό τον κίνδυνο θα πρέπει να συζητήσουμε, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί κοιτώντα τα χρήματα, τα κονδύλια που θα δαπανηθούν ακόμα και όταν το Ταμείο Εξυγίανσης φτάσει στο επιθυμητό και προτινόμενο επίπεδο, αν ρωτιόμαστε, θα αρκέσει να επιλύσει μια μελλοντική Lehman Brothers. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αυτό. Υπάρχει και ένας κίνδυνος ό,τι αφορά την καλή θέληση, αν θέλετε. Μάλιστα, τώρα κατάλαβα το ερώτημά σα. Καταρχά είμαι επίτροπο εσωτερικής αγοράς, Επομένω, όλε τι νομοθεσίε που παρουσιάζω και ο κύριος Φάμπ είναι και στην αίθουσα και αυτός δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα στα πλαίσια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς για διάφορες άλλες πτυχές ε, του χαρτοφυλακίου μου προσπαθώ πραγματικά να δημιουργήσω ένα μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωση της ενιαίας αυτής αγοράς. Και θέλουμε πραγματικά ένα ενιαίο εγχειρίδιο αγορών, μια ενιαία εσωτερική αγορά. Δεν είναι τυχαίο το ότι τονίζω τον όρο αυτό single, ενιαίο και πραγματικά θέλουμε το ίδιο και για την εποπτεία της Τραπεζικής Ένωσης και για το σύστημα εξυγίανσης. Να είναι το σύστημά μας ανοιχτό προς τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν ανήκουν ακόμα στην Ευρωζώνη. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μην δημιουργηθεί αυτή η δυτή νοοτροπία των υπάρχουν δύο ουσιαστικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό όχι για να καθησυχάσω τόσο, όσο για να εξηγήσω το ότι θα έχουμε την ίδια βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία εξυγίανση, η οποία έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να ψηφιστεί, βασίζεται στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Υπάρχει μία ενιαία δέσμη κανόνων, κοινή για όλους, πρώτον αυτόν και δεύτερον έρχομαι στο άλλο σας ερώτημα κύριε Αγαπητέ συνάδελφε, όσον αφορά τα ανασταλτικά μέσα, τους ανασταλτικούς μηχανισμούς που πρέπει να προβλεφθούν, και γι' αυτό το λόγο είπα ότι και οι παρατηρήσεις Άσμουσεν είναι ενδιαφέρουσες, Προκειμένου να έχουμε το σύστημα αυτό των ανασταλτικών μηχανισμών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε και ένα κοινό σύστημα διάσωσης, το οποίο δεν θα στηρίζεται πλέον στα χρήματα των φορολογουμένων. Σαφώς λοιπόν δεν θέλω να δημιουργήσουμε δύο συστήματα, δύο νοτροπίες εξυγένσης. Θα έχουμε μια κοινή ρυθμιστική βάση, η οποία θα εφαρμόζεται με τρόπο συνεκτικό, πιο ομοσπονδιακό αν θέλετε, στην Ευρωζώνη, αλλά οι ίδιοι πάλι κανόνες θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται και εκτός Ευρωζώνης. Νομίζω λοιπόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την ύπαρξη αυτή, την γένεση δύο συστημάτων. Είπατε επίση ότι ενδεχομένω ε, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μην έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση στο νέο Ταμείο Εξυγίανσης. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλε τι ιδέε που έχουν υποβληθεί επιτάπητος αυτή τη στιγμή για να δούμε πώ μπορούμε να προσελκύσουμε εξωτερικό δανεισμό, εξωτερική χρηματοδότηση για το Ταμείο αυτό, αν αυτό κρυθεί αναγκαίο. Ο κύριο Ντομένιτς έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, Προχωράμε σιγά σιγά προς το τέλος της θητείας μας και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό. Εγώ εκτίμησα όλους ιδιαιτέρως και εκτιμώ πάντα το έργο σας. Η άποψή μου πάντως είναι ότι αν χωρίσουμε το έργο σας αυτό σε δύο μεγάλα κεφάλαια, μεταρρύθμιση και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και από την άλλη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, ενδεχομένως να πούμε ότι θα καταφέρουμε να είμαστε πιο ικανοποιημένοι για το πρώτο αυτό κεφάλαιο και όχι τόσο για το δεύτερο. Ποια είναι η δική σας η άποψη σε σχέση με αυτό, δηλαδή σε σχέση με τις προσδοκίες τις δικές σας και σε σχέση με τις απαιτήσει που είχατε. Τι ποσοστό ικανοποίηση έχετε εσεί αυτή τη στιγμή, είστε ικανοποιημένο κατά 60%, κατά 70% σε σχέση με τι αρχικέ σα προθέσει, και τι έχει να μα πείτε σε σχέση με του στόχου που δεν έχουμε ακόμα επιτύχει. Πιστεύετε ρεαλιστικά ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου αυτού, όπω για παράδειγμα η νομοθετική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν θα καταφέρετε να μα δώσετε κάποια περισσότερα δεδομένα όσον αφορά την πραγματική διάρθρωση των τραπεζών και τι συνέχεια μπορεί να δοθεί στην έκθεση Λέκανεν και όσον αφορά το ποσοστό αυτό που δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Πώς επηρεάζει το γεγονός ε, το ότι το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά ε, εμπόδισαν, τροχοπέδισαν τη δική σας ε, την εργασία, τις δικές σας προσπάθειας. προσπάθειες. Κύριε Αν μιλούμε για τους καταναλωτές, ε, για τους πολίτες, που μερικές φορές ε, και ακουσίως χρειάστηκε να σπεύσουν για να διασώσουν τον τραπεζικό τομέα την τελευταία πενταετία σε πολλές χώρες. Όλα αυτά που κάνουμε από κοινού για να εδραιώσουμε τον τραπεζικό τομέα και να το κάνουμε πιο ανθεκτικό χάρη στην εξηγήση, ώστε την χρηματοδοτούν οι ίδιες οι τράπεζες, να γίνει, υπάρχει καλύτερη εποπτεία, καλύτερη ανακεφαλαίωση, περιπτώσεις πτώχευσης να είναι πιο περιορισμένες και σε περίπτωση πτώχευσης ε, να μην πληρώνουν τα σπασμένα οι φορολογούμενοι. Όλα αυτά τα κάνουμε για τους πολίτες. Όπως και το γεγονός ότι αν οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να είναι τόσο ασταθείς ε, ε, και ευμετάβλητες και μερικές φορές στηρίζονται σε αθρές βάσεις, όλα θα πάνε στραβά. Και η μάχη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα θα κερδιθεί με προσπάθειες από όλους και από όλες τις χώρες. Αλλά ποια είναι η βάση, είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σε όλη την περίοδο της κρίσης από την πτώση της ε, Lehman Brothers διαπιστώσαμε ότι η κρίση γονάτισε την ανάπτυξη στην Ευρώπη ή επιδίνωσε την, το, το δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα κτλ. Και, και μετά την απόφαση της 29ης Ιουνίου του 2012, του 2012. Προσπαθούμε αργά αλλά σταθερά να βάλουμε τα θεμέλια και για την Τραπεζική Ένωση είναι για να αποκαταστήσουμε μια σταθερότητα και μια νυφαλιότητα για να προσελκύσουμε τους ε, επενδυτές. Δηλαδή, για πολλούς λόγους μερικές φορές ε, δεν κινούνται οι επενδυτές, αλλά σίγουρα χρειάζονται σταθερότητα, προβλεψιμότητα και θέλουμε να σταθεροποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, και οι επιχειρήσεις, τα εξωτερικά ταμεία, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια κανονιστική σταθερότητα και μια προβλεψιμότητα και διαφάνεια. Και πολλά κείμενα βρίσκονται επιτάπητος, κύριε Ντομένιτσι, υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμβάλλουν σε αυτήν ε, ε, τη βοήθεια και την εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών. Το πακέτο για τους καταναλωτές ε, ή το βασικό κώδικα της τράπεζας, το θέμα της κινητικότητας από τη μία ή την άλλη τράπεζα, τα PRIPS, με την προστασία των καταναλωτών ε, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα θέματα διαμεσολάβησης ε, στις ασφαλίσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα θέματα άμεσα επηρεάζουν και ενδιαφέρουν ε, τον Ευρωπαίο πολίτη και δείχνουν πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του. Και θα ήθελα όλα αυτά τα ζητήματα να διεκπαιρεωθούν και μάλιστα ή δυνατόν πριν το τέλος της χρονιάς αυτής. Τάισεν, e η κυρία Τάισεν από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει την ποιότητα των ισολογισμών των τραπεζικών και αυτό το συζητήσαμε με διάφορους συναδέλφους ήδη σήμερα. Αυτό που αναρωτιέμαι, ο τραπεζικός τομέας ξέρει τι τον περιμένει. Ελπίζω δηλαδή ότι ξέρετε ότι τον περιμένει τραπεζικό τομέα, αλλά βλέποντα τι αντιδράσει ε, στον τύπο, στα μέσα ενημέρωση και βλέποντα και το τι ρωτάει ο κόσμο, αναρωτιέμαι μήπω ήταν χρήσιμο πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει αυτά τα stress test ε, να υπάρξει μια καλή ενημέρωση και προ τον τύπο και προ τα μέσα ενημέρωση για να ενημερώσουμε ότι τα πρότυπα θα γίνουν πιο αυστηρά και άρα να μην ε, φανεί στην πρώτη αφορμή ότι θα ξεσπάσει πανικός και ότι ο κόσμος θα πιστέψει ότι θα ξεκινήσει από την αρχή η πάλι κρίση. Αυτό λίγο με φοβίζει με το πρώτο δηλαδή πρόβλημα που θα ανακύψει να υπάρξει, να ξεσπάσει πανικός. Να μπορέσουμε δηλαδή να μεταφέρουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα έχουν διαμορφωθεί πιο αυστηρά πρότυπα σε ό,τι αφορά τις τράπεζες που θα πρέπει να πληρούν πιο αυστηρά πρότυπα, πιο αυστηρές ε, κανόνες εποπτείας. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω, αν το, δεν νομίζω να το απαντήσετε συγκεκριμένα Μπορεί να, το, να μην το άκουσα. Αλλά πότε θεωρείτε, επιτρέπε ότι θα κάνετε μια συγκεκριμένη πρόταση για την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Ξέρω ότι εργάζεστε από αυτού, αλλά προς το παρόν κάθε κράτος μέλος ετοιμάζει τέτοιες ε, νομοθετικές προτάσεις. Ε, γιατί στην δική μου χώρα, στο Βέλγιο, προβλέπεται από την κυβερνητική συμφωνία ότι θα πρέπει να κατατεθεί σχετική πρόταση. Σε περίπτωση που δεν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κράτου μέλου, σε Βελγίου δηλαδή. Κατά τρίτον, είναι πολύ πρόημο να μιλάμε για δάφνες και απολογισμούς, γιατί έχουμε ακόμα 8 μήνες, αλλά μας δώσατε ένα φυλάδιο για το τι έχει συμβεί. Και αυτό πραγματικά το εξηγώ στον κόσμο. Αλλά κοιτώντας ε, το τι ο τύπος την προηγούμενη εβδομάδα ε, προβάλλει προς τον κόσμο με την πρέτη επέτειο της Lehman Brothers είναι σαν να μην ξέρει ο κόσμος το τι έχει συμβεί σε επίπεδο νομοθετικό σου, τι έχει αλλάξει, ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να τονίσουμε δηλαδή ότι όλα αυτά φυσικά θα γίνουν βήμα-βήμα, ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, αλλά θα πρέπει να γίνει πολύ πιο καλή ενημέρωση, γιατί ο κόσμος πραγματικά λαμβάνει λανθασμένα μηνύματα. Πραγματικά όλη την προηγούμενη εβδομάδα μου με σταματούσε και μου έλεγε ο κόσμος ότι μα δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από, το, από τις ΗΠΑ. Μα τι κάνεις αυτό το κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι έχει συμβεί και το ποια είναι η προπτική μας κυρίως. Ε, ε Κυρία Τάισεν, Θα ήθελα να συνδέσω την πρώτη και την τρίτη ερώτησή σας, γιατί αναφερθήκατε στην επικοινωνία, στην ενημέρωση. Ναι, ως προς αυτό, πιστεύω ότι το quality review όσον αφορά επίσης και τα stress tests που θα ξεκινήσουν ε, το 2014, το νέο κύμα δηλαδή των stress tests, νομίζω ότι ως προς αυτά θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα στοιχεία αυτά στα πλαίσια μιας παγκόσμιας σφαιρικής στρατηγικής. Και αυτό ακριβώς είπα και στους υπουργούς που συνάντησα το Σάββατο το πρωί. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Τους είπα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, σημα... πάρα πολύ προσεκτικοί με την ενημέρωση και την επικοινωνία και ότι θα πρέπει το security review της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να γίνει με έναν τρόπο εντελώς ανοιχτό και ότι κατά αυτόν τον τρόπο επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε και όλες τις δραστηριότητες της CBA όσον αφορά τα δοκιμαστικά τεστ για τις τράπεζες. Ότι θα πρέπει με ένα σοβαρό τρόπο να επιτελέσουμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά να ενημερώσουμε κατάλληλα και τους πολίτες και να αποφύγουμε οποιαδήποτε επιθανολογία όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών των ενεργειών. Έχω ενημερώσει λοιπόν όλους τους υπουργούς οι οποίοι εργάζονται στον τομέα αυτό και τους είπα ότι θα πρέπει να επιτελέσουν παράλληλα και αυτό το στρατηγικό έργο της επικοινωνίας, της πληροφόρησης. Και δεν είμαι μόνος, κύριε Τάισεν, που λέω τα πράγματα αυτά. Όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στο στρατηγικό αυτό έργο και επιθυμεί να καταστήσει το έργο αυτό κατανοητό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Όσον αφορά την, την ανάταξη των τραπεζών, την ανδιάρθρωση των τραπεζών, θα υποβάλω μια πρόταση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο. Ουσιαστικά οι ίδιες ομάδες εργάζονται και για το ζήτημα αυτό δεν πρόκειται να σας πω αυτή τη στιγμή κάτι διαφορετικό. Έχω πολύ ε, έμπειρους ε, και ικανούς συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με απόλυτη σοβαρότητα και ανάλωσαν όλο το καλοκαίρι προκειμένου να εργαστούν για το ζήτημα αυτό της ε, Τραπεζικής Ένωσης, της Τραπεζικής εξυγίανσης και ασχολούνται προφανώς και με την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Εθνικά ορισμένα κράτη-μέλη κινούνται παράλληλα, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, που καταρτίζουν τα δικά τους σχέδια, τα οποία όμως δεν αποκλείουν πολύ μεταξύ τους. Ξέρω ότι και οι Άγγλοι έχουν κάνει κάτι ανάλογο μέσω των εργασιών του κυρίου Βίκερς. Ε, υπέβαλαν και αυτή μία πρόταση. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να ισχύει. Πάντως, εγώ έδωσα πρωταρχική προτεραιότητα σε όλες τις οριζόντιες προτάσεις είτε αναφερόμαστε στην ανακεφαλαιοποίηση, στη διακυβέρνηση, την εποπτεία, την εξυγίανση, όλους αυτούς τους τομείς που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας, της διαφάνειας, της προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών, των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Αρκεί όμως αυτό. Η απάντηση είναι όχι. Είμαι πεισμένος ότι πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και να καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τη διαχείριση των κινδύνων, ιδίως όσον αφορά το property trading, το οποίο παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα, το market making, το οποίο πρέπει να αποσαφινιστεί. Επεξεργαζόμαστε πάντως τα ζητήματα αυτά και θα σας παρουσιάσω τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέλλον θα γίνει μια πρώτη εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο των Υπουργών. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εγκριθούν τα κείμενα αυτά και είναι σημαντικό τα αντίστοιχα εθνικά κείμενα που υπάρχουν να μπορούν να συνδυαστούν με τις ευρωπαϊκές αυτές προτάσεις. Τέλος, κυρία Τάισεν, αναφερθήκατε στο ζήτημα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης. Ουδέποτε εγώ ζήτησα από δημοσιογράφους ή από παρατηρητές να είναι ποιικείς μαζί μου ή συγκαταβατικοί. Και ξέρετε ότι εδώ και τρία χρόνια, μάλιστα στις 10 Φεβρουαρίου του 2010, είπα ότι θέλω πραγματικά να αξιολογηθώ βάσει τις δράσης την οποία αναλάμβανα τη στιγμή εκείνη. Και ο Ευρωπαίος πολίτης, στον οποίο αναφερθήκατε, στον οποίο πραγματικά εμεί πρέπει να λογοδοτήσουμε και εσείς και εγώ, ο Ευρωπαίος λοιπόν πολίτης τι βλέπει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι βλέπει την αλήθεια την οποία εξέφρασα και εγώ στην εισαγωγική μου ομιλία, ότι οι περισσότεροι νόμοι οι οποίοι έχουν πλέον εγκριθεί, οι περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες για τις οποίες καταβάλαμε τόσο πολλές προσπάθειες, τελικά εγκρίθηκαν και στην καλύτερη των περιπτώσεων οι περισσότεροι όμως αυτοί νόμοι δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν ακόμα 3,5 χρόνια μετά την έναρξη των προσπαθειών μας, μολονότι εμείς αρχίσαμε να εργαζόμαστε πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Το ίδιο ισχύει και για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ξέρετε ότι αντίστοιχες αμερικανικές νομοθεσίες παρουσιάζουν ε, την ίδια πολυπλοκότητα και ακόμα δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να εργαστούμε πιο γρήγορα, δεν νομίζω. Πρέπει να τηρήσουμε τον χρόνο τη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να πούμε την αλήθεια προ τον Ευρωπαίο πολίτη, ότι απαιτείται χρόνο. Πάντω, το έτος αυτό είναι ένα έτος κλειδί, γιατί οι περισσότερες από αυτές νομοθεσίες στα τέλη του 2013, στα αρχές του 2014, θα αρχίσουν επιτέλους να ισχύουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα αλλάξει ριζικά τραπεζικός τομέα όσον αφορά την εποπτεία, όσον αφορά την εξυγίανση. Όπως έχει ήδη συμβεί με τις εταιρείε επιστολεπτικής αξιολόγησης, όπως θα γίνει αργότερα το 2014 με άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανυπομονούν να δουν αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή, νομίζω όμως ότι αν καταβάλουμε τις κατάλληλες προσπάθειες εξήγησης και πληροφόρησης, σωστής ενημέρωσης, θα καταφέρουμε να τους, κάνουμε, να τους κάνουν να καταλάβουν πώς έχουν τα πράγματα. Επίσης, είναι σημαντικό να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε και σε κάποια ζητήματα τα οποία πραγματικά γίνονται πιο κατανοητά ή αφορούν πιο άμεσα από τον Ευρωπαίο πολίτη στην καθημερινή του ζωή. Το να καταφέρνει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα, νομοθετήματα τα οποία έχουμε εγκρίνει και τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα ως Ευρωπαίους πολίτες. Κυρία Φερέρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας και για την αιμονή σας και την επιμονή σας να διεκπαιρεώσετε εγκαίρως σε αυτό το πρόγραμμα. Και μπορείτε να υπολογίζετε όπως έγινε μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα σταθεί στο πλευρό σας όπως στάθηκε. Έχω μερικές ερωτήσεις. Καταρχήν για την Τραπεζική Ένωση. Η πρώτη μου ερώτηση έχει μεθοδολογικό χαρακτήρα. Στο κείμενο για την ενιαία εξυγίαση περιλάβατε και πολλά στοιχεία από την οδηγία RRD για την ανάκαμψη και την εξυγίαση. Υιοθετήσατε όμως την ε, εκδοχή του Συμβουλίου τι σημαίνει αυτό, ότι κάποια στοιχεία της πρότασης του Συμβουλίου κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία για τον ε, νέο μηχανισμό εξυγίασης ή όλα μένουν ανοιχτά από τη στιγμή που συνεχίζεται ακόμη ο τριμερής διάλογος μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα το θέμα του bailing το 8%. Και μία ακόμη ερώτηση που είναι περισσότερο σχόλιο. Όταν η εξυγίαση περάσει στο κοινοτικό επίπεδο, υπάρχει σύγκληση των απόψεων ότι χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό backstop, ένα ευρωπαϊκό ανασταλτικό μηχανισμό. Και θα θέλαμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε, αλλά σε αρμονία με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και όχι διάσταση. Επίσης, μία διάρθρωση που χρειάζεται για το Συμβούλιο, για το Διοικητικό Συμβούλιο και μία διαχωρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες Επιτροπής και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Board, του Συμβουλίου αυτού και πού θα, όταν χρειάζονται συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις για την εξυγίανση προβλέπετε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ή τις Εθνικές Αρχές Εξυγίασης, ώστε αυτό το Συμβούλιο, αυτό το σώμα να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έργο του. Ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτού της νομοθετικής πρότασης είναι η τις εθνικες αρχες εξυγιασης ωστε αυτο το συμβουλιο αυτο το σωμα να μπορεσει να ανταπεξελθει στο εργο του ενας απο τους λογους υπαρξης αυτης της νομοθετικης προτασης ειναι η προστασια των καταθετών. Πιστεύω ότι υπάρχει δυναμικό για την προστασία των καταθετών με βάση αυτή την νομοθετική πρόταση. Κυρίως όμως ε, όταν ε, μιλούμε για το σύστημα εγγύης καταθέσεων που θα συμβάλλουν στο θέμα της εξήγησης, δηλαδή τα DGS να περάσει στο bail-in. Αλλιώς δεν θα απομακρυνθούμε από τα γνωστά περιστατικά του FDIC στις Ηνωμένε Πολιτείες ή το Institutional Protection Scheme σε περίπτωση κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι υπάρχουν βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στην τρέχουσα νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Φερέιρα για τα σχόλιά σας, ε, για το κοινό μας έργο. Ναι, στο κείμενο για την Τραπεζική Ένωση και την εξυγίανση, το SRM, έβαλα και ένα τμήμα από το κείμενο του Συμβουλίου, από την κοινή πολιτική θέση του Συμβουλίου, που ήταν το απάβγασμα πολύ ωραίων συζητήσεων και ολονύκτιων μερικές φορές. Για νομικοτεχνικούς λόγους το έκανα αυτό κυρία Φεραίρα. Πάντως η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Η πρόταση αυτή δεν ε, προδικάζει την ε, δημοκρατική έκβαση αυτών των συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εξυγίασης. Το έκανα για νομικοτεχνικούς λόγους, αλλά δεν προδικάζει τίποτα σε ό,τι αφορά την πορεία των συζητήσεων. Δεύτερον, για το backstop, τον ανασταλτικό αυτομηχανισμό. Εγώ σας πρότεινα, εισακούγοντας το Κοινοβούλιο, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίασης στο επίπεδο της Ευρωζώνης, ένα είδος δηλαδή ανασταλτικού μηχανισμού ιδιωτικού, γιατί ε, ο μηχανισμός αυτός, ε, το ταμείο αυτός χρηματοδοτείται από τις τράπεζες και έχουμε και ένα δημόσιο ανασταλτικό μηχανισμό που λειτουργεί σήμερα και θα λειτουργήσει με εσωτερικές μεθόδους απόφασης που είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Αυτά ως προς τους τρόπους που έχουμε προβλέψει για τη χρήση την επέμβαση αυτών των ανασταλτικών μηχανισμών. Που πραγματικά όμως θα είναι ίστατη λύση σε ακραίες περιπτώσεις. Γιατί όλο αυτό το νομοθετικό πλωστάσιο που εφαρμόζουμε έχει στόχο ότι καλύτερα ανεκεφαλοποιημένε και καλύτερα δικούμενες τράπεζες δεν θα βρεθούν ε, σε, καμία περίπτωση σε κατάσταση πτώχευσης. Αν τώρα για σε λόγους συγκυρίας ε, ε, διαφόρων φουσκών δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει φυσικά να χρησιμοποιήσουμε το νομοθετικό πλωστάσιο που προβλέπει πρώτα το bail-in δηλαδή την παρέμβαση των μετόχων και των πιστωτών που αναλαμβάνουν τη διάσωση και στη συνέχεια τους υπόλοιπους ανασταλτικούς μηχανισμούς, στους οποίους προσφεύγουμε με τη σειρά που ανέφερα, πρώτα ιδιωτικούς, μετά δημόσιο. Πάντως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ακριβώς για να έχουμε ε, όσο λιγότερη ανάγκη γίνεται αυτών των μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά το θέμα των, της Επιτροπής, ε, του Συμβούλιο ήταν κατά, ε, ακούστηκαν πολλές επιφυλάξεις από το Συμβούλιο για το ρόλο που πρότεινα εγώ για την Επιτροπή. Βέβαια, εγώ είπα ότι δεν θα είναι η Επιτροπή η αρχή εξυγίαση. Ούτε διεκδικούμε κα... κάποιον τέτοιο ρόλο. Ακόμη και αν έχουμε εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, γιατί η πολιτική των κρατικών ενισχύσεων ε, ε, μα ενδιαφέρει και συνεχίζουμε το ρόλο μα, ειδικά με τον νέο κανονισμό που πρότεινε ο κύριος Σαλμούνια για την αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων ε, στον τραπεζικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να παίξει το ρόλο μιας αρχής εξηγίασης. Χρειαζόμαστε όμως ένα θεσμικό όργανο που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, που θα πρέπει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό. Και σκέφτηκα, ποιο είναι, ποιο είναι τα όργανα που έχουν δυνατότητα άμεσης δράσης. Γι' αυτό πρότεινα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θεωρούσε ήταν ε, το μη χείρο στην περίπτωση αυτή. Και είπα τους στους υπουργού, αν έχετε καμιά καλύτερη ιδέα, να μας την υποβάλλετε και θα την εξετάσουμε αντικειμενικά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό, θα πατήσει το κουμπί και θα ξεκινήσει ένα σχέδιο εξυγίανση που έχει γίνει από το Συμβούλιο Εξυγίανση από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες, γιατί η οδηγία προβλέπει κάθε τράπεζα να ετοιμάσει το σχέδιο εξυγίανση της. Αν χρειαστεί τελικά αυτή η εξυγίαση, όταν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η ΕΚΤ, το board, το συμβούλιο αυτό, θα ετοιμάσει την οργάνωση της εξυγίασης, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πατήσει το κουμπί και μετά το Συμβούλιο Εξυγίασης, αυτό το board θα εφαρμόσει την εξυγίαση σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Αυτά προβλέπουν οι προτάσεις. Βέβαια όλα, είναι, όλα βρίσκονται να εξελίξει ανάλογα με τις συζητήσεις που θα έχουμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεταχείριση των καταθετών, αυτό είναι από τα πιο ευαίσθητα και περίπλοκα θέματα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το είδαμε και με την κρίση στην Κύπρο. Εκεί ένα επικοινωνιακό λάθος δημιούργησε τεράστια φόρτιση και συναισθηματικές αντιδράσεις και φυσικά μέχρι 100.000 θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση καταθέσεων και εμείς προτιμήσαμε τους καταθέτες ε, με βάση την προσέγγιση του Συμβουλίου. Θα συνεχιστεί φυσικά ο τριμερής διάλογος και είναι ένα θέμα στο οποίο δραστηριοποιείται ο κύριος Σάιμον. Θα έχουμε εγγύηση καταθέσεων ε, αποτελεσματική. Ένα σημείο που δεν έχει ακόμη διεκπαιρεωθεί. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις Πάντως θέλουμε οι εγγύσεις να είναι αποτελεσματικές και τα κονδύλια που θα προβλέψουμε για αυτές αξιόπιστα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε, έχουμε χρόνο. Τέσσερι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και 20 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μα. Ο κ. Φαμπρίτσιο Δάζο από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε, το λόγο που εκφώνησε στην αρχή της συνεδρίασής μας και τον ευχαριστώ επίσης και για τον οδικό χάρτη στον οποίο αναφέρθηκε που είχε ως στόχο την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, την εποπτεία τους επίσης, πώς μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές, σε αυτούς οι οποίοι ως ιδιώτες τελικά χρησιμοποιούν τα χρήματά τους προκειμένου να κάνουν επενδύσεις μέσω του τραπεζικού μας κλάδου. Νομίζω λοιπόν ότι Συναντήσατε αρκετές δυσκολίες στις προσπάθειές σας και νομίζω ότι το πιο δύσκολο θα ήταν ε, έργο ενδεχομένω το να ήταν κανείς επίτροπος ασφάλειας, ναυτιλιακής ασφάλειας μετά την βήθηση του Τιτανικού. Μόνο αυτό θα είχε πιο δύσκολο έργο από εσά. Είπατε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο, κάτι στο οποίο εσείς λίγο αναφερθήκατε στο λόγο σας, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο. Θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να αρχίσει να συγκλίνει όλο και περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Εσείς τι πιστεύετε όσον αφορά μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση από δημοσιονομικής πλευράς ή από φορολογικής πλευράς, αν υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα να μην φορολογούνται μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες από, συγκεκριμένους, από συγκεκριμένες μεθόδους χρηματοδότησης, ιδίως από τη χρηματοδότηση εκείνη η οποία επιφέρει πραγματικά μια σημαντική προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εσείς νομίζω ότι αναφερθήκατε στο λόγο σας στην σύγκληση αυτή που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο τραπεζικό τομέα και τις ανάγκες πραγματικής οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπατε ότι αυτό θα μπορέσει να αποτελήσει τη βάση μιας σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να επιλύσουμε την μεγάλη αυτή δεύτερη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή πέρα από τη χρηματοπιστωτική κρίση έχουμε και την οικονομική και κοινωνική κρίση που ακολουθεί. Κύριε Μπερτότα. Σας ευχαριστώ επίσης για τα όσα είπατε για την εργασία που από κοινού έχουμε κάνει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αναφερθήκατε επίσης στον Τιτανικό. Είναι σαφές ότι πριν από 2,5 χρόνια παραλίγο να εκτροχιαστεί ο σιδηρόδρομος του Ευρώ, να το θέσω έτσι εξαιτία τη οικονομική κρίση, η οποία προήλθε από τι Ηνωμένε Πολιτείε, εξαιτία των αδύναμων χαρακτηριστικών των τραπεζών σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, εξαιτία τη κακή διασύνδεση που υπήρχε μεταξύ του τραπεζικού χρέου και του δημόσιου χρέου, επίση ε, εξαιτία ενό πολύ υψηλού επίπεδου δημοσίου χρέου, εξαιτία μια ε, μη ικανοποιητική διακυβέρνηση τη Ευρωζώνη, μολονότι είχε κάνει πολλέ εξαγγελίε ο Ζακ Ντελόρ πριν από πάρα πολλά χρόνια προ αυτό, εξαιτία όλων αυτών των λόγων παραλίγο να εκτροχιαστεί το τρένο. Και δεν έγινε βέβαια κάτι αυτό χάρη στην έγκαιρη ε, δράση της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χάρη στην έγκαιρη δράση πολλών δεξιών και αριστερών κυβερνήσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε όλοι από κοινού να βάλουμε τα πράγματα πάλι στο σωστό τους πλαίσιο. Καταφέραμε να κάνουμε τις ράγες του τρένου να είναι παράλληλες και να μην αποκλίνουν και βλέπουμε ότι το τρένο, και χρησιμοποιώ ακόμα την ίδια εικόνα, αρχίζει σιγά σιγά να επανακινείται και βλέπουμε ότι έχει επανέλθει μια κάποια ηρεμία. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα και επαγρύπνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταξίδι μας αυτό, για να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, των Ευρωπαίων επενδυτών, καθώς επίσης και των αγορών, θα πρέπει πραγματικά να υλοποιήσουμε τα όσα λέμε και θα πρέπει τα όσα λέμε να λειτουργούν στην πράξη, να λειτουργούν αποτελεσματικά και αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που καταβάλουν προσπάθειε για να ελέγξουν το χρέο του. Ο συνάδελφό μου, Όλη Ρεν, καταβάλει προσπάθειε προκειμένου να υπάρχει η ο κατάλληλο δημοσιονομικό συντονισμό και εξυγίαση στα κράτη-μέλη. Εγώ προσπαθώ από την άλλη να έχουμε μια οριζόντια ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από όλα αυτά όμω, θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε και την οικονομική ανάπτυξη, να μην βαρύνουμε τις επενδύσεις με μια έντονη γραφειοκρατία, θα πρέπει να προωθήσουμε σωστά τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Αναφερθήκατε επίσης στην ερώτησή σας και σε κάτι ακόμα το αν θα μπορούσαμε να απαλλάξουμε φορολογικά κάποια έσοδα επιχειρήσεων και κάποια έσοδα τα οποία προέρχονται από τις αγορές. Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε, αλλά πρέπει να πούμε ότι στα πλαίσια του φυστάμενου δικαίου Όποιο φορολογικό μέτρο και αν λαμβάνεται αυτή τη στιγμή είναι εθνική αρμοδιότητα. Κάθε φορά προσπαθούμε να συντονίσουμε τα φορολογικά μας συστήματα, όπως ο Επίτροπος Εμέτα προσπαθεί να κάνει πολλές φορές, με πολύ κουράγιο μάλιστα, γιατί ξέρω ότι εγώ ως Επίτροπο εσωτερική Αγοράς δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έχουμε ή ότι έχουμε 28 διαφορετικές φορολογικές βάσεις για τις εταιρείε, 28 διαφορετικές εταιρικές φορολογικές βάσεις σε μια εσωτερική αγορά. Έχουμε μάλιστα και μια οικολογική φορολογία μία πλούστευση που προσπαθούμε να προωθήσουμε όσον αφορά το φόρο τη προς φέμενης αξίας, βλέπω ότι προχωράμε πάρα πολύ αργά. Ακριβώς επειδή για τα ζητήματα αυτά απαιτείται απόλυτη ομοφωνία. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να προσπεράσουμε το εμπόδιο αυτό της ομοφωνίας και να ζητήσουμε και για το φορολογικό τομέα, για κάποιες πτυχές του τουλάχιστον, μία ενισχυμένη συνεργασία για τις χώρες εκείνες οι οποίες επιθυμούν να συγκλίνουν πιο γρήγορα στα πλαίσια της Ευρωζώνης βέβαια κυρίως. Τι κάνουμε τώρα εμείς όμως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από νομοθετικής πλευράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που κάνω εγώ με τον Επίτροπο Ταγιάννη σε πολλούς τομείς είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε μια κάποια διαφοροποίηση αν μη τι άλλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να υπάρχει ένα ξεχωριστό καθεστώς για αυτές όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα, όσον αφορά τη διαφάνεια όσον αφορά το CRD4, να καταφέρουμε δηλαδή να ενισχύσουμε περισσότερο τις τράπεζες εκείνες οι οποίες δανειοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είμαστε λιγότερο αυστηροί, να έχουμε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για τις τράπεζες αυτές, οι οποίες χρηματοδοτικά ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να διαφοροποιήσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην εξαρτώνται μόνο από τις τράπεζες, αλλά μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα χρηματιστήρια. Και για αυτό το λόγο θέλω να προωθήσω ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξεκίνησε και μια όλη εργασία για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Στα πλαίσια της πρότασης αυτής λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό, ε, ένας ευρωπαϊκός αποτεμευτικός λογαριασμός για ποιο λόγο να μην φανταστούμε ότι σε μερικά χρόνια θα καταφέρουμε να έχουμε ένα εγγυημένο ευρωπαϊκό προϊόν όπου η ιδιωτική αποταμίευση θα μπορούσε να συλλεχθεί και να νίκει τελικά σε ένα ευρωπαϊκό αποταμιευτικό λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι τέτοια προδραστικά μέτρα πρέπει να προωθήσουμε. Ε, Μάλιστα, έχουμε τρεις ερωτήσεις. Κύριο Σάντζες Πρεσέντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και κρίνω πολύ θετικά τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ θετικές και οι πρωτοβουλίες και η στάση που κράτησε ο Επίτροπος ως προς τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση. Εγώ θα επικεντρωθώ τώρα στα σημεία που χρήζουν συμπλήρωση και βελτίωση γιατί Υπάρχει κολλησιεργία σε ορισμένα θέματα και εκκρεμότητε. Ε, για την ενυπόθηκη πίστη, τα στεγαστικά δάνεια. Ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έμεινε εκκρεμέ ένα τεχνικό θέμα ω προ την εφαρμογή τη οδηγία. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεκπαιρεώσει το θέμα σε πρώτη ανάγνωση θα ήταν πραγματικά τραυματική εμπειρία να έχουμε καταλήξει στη συμφωνία ω προ την ουσία και για ένα τεχνικό θέμα που έμεινε εκρεμές να μην καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα σε πρώτη ανάγνωση. Μήπως έχετε κάποιε πληροφορίες για αυτή την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Ό,τι αφορά την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη θέλουμε να ενισχύσουμε τη... τα υπεύθυνα στεγαστικά δάνεια. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την χρέωση, την ιδιωτική χρέωση, τα, χρέη των οικοκυριών. Και ξέρω ότι η υπεύθυνη, ο υπεύθυνο δανεισμό δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στου καταναλωτέ, γιατί είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στου καταναλωτέ. Καλό θα ήταν να ε, αναφερθούμε και σε άλλε πτυχέ. Σε ό,τι αφορά την ε, διαρθρωτική μακροοικονομική μεταρρύθμιση. Ήδη έχει αναγγελθεί η πρωτοβουλία για το φθινόπωρο και θα ήθελα να μου πείτε πώς θα συνδυάσετε αυτές τις αναγκές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση με το σύστημα της Οικουμενικής Τράπεζας ε, που έχει λειτουργήσει στην Ευρώπη. Κύριε Πρεσέδο, με χαροποίησε ιδιαίτερη έκβαση της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ θερμά. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε ε, σε, ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς να έχουμε νέο πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια, αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Βέβαια, έμεινε κρεμές ένα θέμα που μας υπενθυμίσατε, τεχνικό, μια διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή της διοργανικής αυτής συμφωνίας. Αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας και τα ε, διευκρινιστικά έγγραφα που απαιτείται. Εγώ ε, κατανοώ τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο να κινηθεί και να βρεθεί μια συμφωνία. Γνωρίζω ότι η πρόεδρό σας, η ε, κυρία Σάρον με την οποία μίλησα, είχε προσωπικές συνομιλίες με τον Λιθουανό Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και την Παρασκευή και το Σάββατο και εγώ συνομίλησα μαζί του για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα αρχή σημαντικό για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν θα μπλοκάρουμε την εφαρμογή του κειμένου για τα ενυπόθηκα δάνεια που είναι πολύ σημαντικά εξαιτίας αυτού του τεχνικού ζητήματο. Θα πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία. Και εγώ διαβεβαίωσα την ε, Λιθανική Προεδρία για την απόλυτη προθυμία μου να διευκολύνω την ε, σύγκληση απόψεων και ανέβρεση λύση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ε, οπότε το, έχουμε στο αυτό το κείμενο για την ενυπόθηκη πίστη και τα ενυπόθηκα δάνεια τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να καταλήξουμε σε υπεύθυνα δάνεια γενικά πέραν του, των προτάσεων για τα στεγαστικά αυτά δάνεια που προτείνουμε στο κείμενο, θέλουμε γενικά οι καταναλωτές χρηματοπιστωτικών προϊόντων, είτε είναι δάνεια είτε άλλα προϊόντα, να τη χάνουν μεγαλύτερου σεβασμού και καλύτερη ε, ενημέρωση για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Αυτό το κάνουμε για όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θέλουμε αυστηρή ενημέρωση του πελάτη για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο πελάτης αυτός ο καταναλωτής. Και αυτό το θέμα εφαρμόζεται σε πολύ περισσότερα ζητήματα πια. Και θέλουμε να υλοποιήσουμε και αυτή την ιδέα των υπεύθυνων δανείων και με το κείμενό μας για τα ενυπόθηκα δάνεια. Η κυρία Λούλινγκ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πριν από μία εβδομάδα περίπου υποβάλλεται μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη ρύθμιση των νομισματικών ταμείων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόταση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο τομέας αυτός βέβαια έχει αντιδράσει, μπορούμε να πούμε, με έναν τρόπο μετριασμένο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θέτει να αφιβόλω την σκαλές προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να γνωρίζω πάντως κύριε Επίτροπε ποιες είναι οι δικές σας αντιδράσεις απέναντι σε αυτούς που λένε ότι οι προτινόμενες αλλαγές τελικά υπερβαίνουν ε, τους υφιστάμενους κανόνες ε, όσον αφορά τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητικές αξίες. Ξέρετε ότι υπάρχει ήδη μία ρύθμιση για τους οργανισμούς αυτούς, μία ρύθμιση η οποία είναι και αρκετά επιτυχής μάλιστα. Στην εφιστάμενη τώρα συγκύρια όσον αφορά των πολύ χαμηλών επιτοκίων, αυτά τα νομισματικά ταμεία αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες και το να επιβάλλουμε επιπλέον πολύ αυστηρούς κανόνες για τα ταμεία αυτά ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει για αυτά την τελεσίδικη καταδίκη τους. Εσείς θέσατε ένα ποσοστό της τάξης του 3% και νομίζω ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν βρίσκει σύμφωνο στους παράγοντες του κλάδου αυτού. Τι πιστεύετε λοιπόν, ποια είναι η δική σας η αντίδραση όσον αφορά τις επικρίσεις του εν λόγω τομέα, όσον αφορά τις δικές σας δηλαδή τις προτάσεις και είστε έτοιμος να αναθεωρήσετε κάποιες από τις προτάσεις σας και ανηγένει. τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να ρυθμίσετε ακόμα περισσότερο έναν τομέα ο οποίος είναι ήδη αρκετά κατακαιρματισμένος και ιδιαίτερα ευάλωτο εξαιτία τη υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να βρείτε μια κάποια πιο εξορροπημένη προσέγγιση. Ο Επίτροπος στον κύριο Σάντσετς Πρεσέντο καταρχάς με την άδειά σας να πω κάτι γιατί ξέχασα να απαντήσω πριν από λίγο στην ε, ερώτησή του όσον αφορά την μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Κύριε Σάντσετς Πρεσέντο, προετοιμάζω την εν λόγω μεταρρύθμιση κάνοντας μια, ένα διαχωρισμό της στάθμισης των κρίσεων με βάση το κινδύνου, με συγχωρείτε, με βάση του έργου που επιτελεί πραγματικά η τράπεζα. Δηλαδή, αν πραγματικά χρηματοδοτεί πελάτε, αν πραγματικά συμβάλλει στην πραγματική οικονομία. Και θέλω πραγματικά να, να σεβαστώ και την διαφορετικότητα στα πλαίσια του τραπεζικού τομέα. Αν δείτε τα διάφορα προβλήματα ή τι κρίσει που έχουμε στο τραπεζικό τομέα, Βλέπουμε ότι έχουμε από τη μια επενδυτικέ τράπεζες όπως οι Lehman Brothers, άλλες μεγάλες τράπεζες ή τράπεζες οι οποίες διαφοροποιούνται σε άλλους τομείς. Έχουμε πολλές διαφορετικές τράπεζες, πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και εγώ ουσιαστικά θα ήθελα μέσω της πρότασής μου να σεβαστούμε αυτή τη διαφορετικότητα η οποία ήδη υπάρχει, την ποικιλία, την ποικιλομορφία που ήδη υπάρχει στο τραπεζικό τομέα, το οποίο είναι κάτι πολύ θετικό για τον τραπεζικό τομέα. Ξέρετε ότι έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες, αλλά έχουμε περίπου και 4 εκατομμύρια μικρότερες τράπεζες. Κυρία Λούλιν τώρα, απαντώντας ε, στο δικό σας το ερώτημα, το Financial Stability Board ουσιαστικά μας ε, ζήτησε να απαγορευθούν ε, τα εναλλακτικά ταμεία και ιδίω αυτά τα οποία ονομάζουμε συνάβα, δηλαδή ταμεία σταθερής αξίας. Αυτό προβλέπεται στο κείμενο. Εγώ ακολούθησα τις τέσσερις μεγάλες συστάσεις του Ιούσκο όσον αφορά το παράλληλο τραπεζικό σύστημα στην ε, εν λόγω πρόταση την οποία επέβαλα. Δεν είπα ότι θα πρέπει να απαγορευτούν αυτά τα ταμεία για δύο λόγους. Πρώτον, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο της σταθερότητας και της ασφάλειας με άλλα μέσα και όχι μέσω της απαγόρευσης. Δηλαδή πρώτα το πετύχουμε αυτό μέσω της χρηστής διακυβέρνησης, μέσω της διαφάνειας, μέσω της σταθερότητας, μέσω αυτής της ε, ζώνης προστασίας του 3% που πρότεινα. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά και όχι την απαγόρευση. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ε, τα ταμεία αυτά ουσιαστικά αποτελούν τη βάση μιας πολύ σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας στο Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Και επομένως τα μέτρα τα οποία πρότεινα πραγματικά λαμβάνουν υπόψη μου τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι προτάσεις μου στις χώρες αυτές. Έτσι λοιπόν όσον αφορά την ε, σταθερή αυτή αξία, η πρόταση που έκανα, την οποία θα συζητείτε εσείς και το Συμβούλιο, είναι να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τα ταμεία αυτά, να υπάρχει αυτή η ζώνη ασφάλειας του 3% που νομίζω ότι είναι ανεκτή για τα ταμεία αυτά, και αν υπήρχε πραγματικά αυτό το περιθώριο ασφάλειας, τότε τα περισσότερα από τα προβλήματα τα οποία είδαμε στο παράλληλο τραπεζικό σύστημα εξαιτίας ε, της κακής κεφαλαιοποίησης των ταμείων αυτών, δεν θα είχαν εμφανιστεί. Τα ταμεία αυτά θα είχαν καταφέρει τελικά να αντέξουν την κρίση. Μιλάμε για κάποια ταμεία τα οποία πειράζουν πάρα πολύ την οικονομία, ξέρετε. Πρόκειται για ταμεία τα οποία αντιστοιχούν σε χίλια δισεκατομμύρια όσον αφορά τις συναλλαγές. Ξέρετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις αυτές όσον αφορά το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και γι' αυτό στις πρώτες μας μάλιστα προτάσεις απευθυνθήκαμε ειδικά, στοχεύσαμε ειδικά τα ταμεία αυτά. Ξέρω ότι ορισμένοι θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ δρακόντια, άλλοι πάλι θεωρούν ότι δεν αρκούν. Εγώ νομίζω ότι έχουμε επιλέξει την μεσαία οδό, δηλαδή να προωθήσουμε περισσότερο τη διαφάνεια. Ο κύριος Ραμόν Τρεμόσα είναι τελευταίος ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελευταία ερώτηση για το ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης των τραπεζών. Κύριε Επίτροπε, διαπιστώνω με ανησυχία ότι πολλές κυβερνήσεις δεν θέλουν να εφοδιάσουν τον ενιαίο αυτό μηχανισμό εξυγένση με αρκετέ αρμοδιότητε για να διαρθρώνει και να εξηγένει τι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή πρόταση ε, ενιαίου μηχανισμού εξυγένση χωρί αλλαγή, προηγούμενη αλλαγή τη συνθήκη. Μπορείτε να δώσετε περισσότερα επιχειρήματα για το σημείο αυτό. Κύριε Τρεμόζη, η απάντησή μου είναι καταφατική. Ναι, πιστεύω με βάση και τη γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας ε, που συνάδηκε με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι είναι δυνατόν να θεσπίσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εξυγίανσης στην Ευρωζώνη με, βάση, με νομική βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης. Και το συζητήσαμε αυτό, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις κυβερνήσεις ε, και νομίζω ότι η νομική αυτή βάση είναι πολύ σταθερή και έγκυρη. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα και προηγουμένως. Σημαίνει ότι θα είναι, οριστικό αυτό, θα είναι οριστική αυτή η λύση, ότι είναι ιδεώδης και δεν επιδέχεται βελτιώσει. Όχι, αλλά θέλουμε να ισχύσει αυτός ο μηχανισμός εξηγήσης το συντομότερο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε δεχόμενο μελλοντική κρίσης και να μπορούμε να οργανώσουμε με ευφύ τρόπο μια συντεταγμένη πτώχευση, αντί να ε, αυτοσχεδιάζουμε τελευταία στιγμή, την τελευταία ώρα, χωρίς προηγούμενη διαδικασία λήψη αποφάσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών. Θέλουμε με την πρόταση αυτή έναν ολοκληρωμένο τρόπο για το bailing και την ε, οδηγία για τη εξυγίαση χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τα σπασμένα ο φορολογούμενος και να εφαρμόσουμε αυτόν τον νέο μηχανισμό εξυγίασης για την Ευρωζώνη. Τώρα, αν τροποποιηθεί η συνθήκη κάτι που είναι ευκταίο σε μεταγενέστερο στάδιο, ε, ιδιαίτερα για διάφορα σημεία λειτουργίας της Ευρωζώνης, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν κάποιες ρυθμίσεις για να βελτιωθεί ο μηχανισμός εξυγίασης. Είπα πριν από λίγο ότι ο μηχανισμός αυτός, ε, ο μηχανισμός ε, σταθερότητας που υπάρχει αλλά είναι διακυβερνητικός και προβλέπει αποφάσεις με ομοφωνία, μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να γίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίαση. Εγώ δεν έχω ιδεολογικά προβλήματα, απλώ θέλω ένα σύστημα που να λειτουργεί εύρυθμα, δεδομένων των προβλημάτων που είχαμε να εξηγένουμε τι ε, ε, τράπεζες τελευταία στιγμή, ήδη στριμωγμένοι στον τοίχο, με ε, εθνικέ αρχέ που δεν είχαν ε, πείρα ούτε προηγούμενη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή συνεννόησης. Θέλουμε ένα σύστημα που θα Ελπίζουμε να λειτουργήσει από το 2014, ας συμφωνήσουν οι κυβερνήσει. Εγώ ευελπιστώ ότι θα ληφθεί απόφαση και φυσικά σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μπορεί το, στοιχείο, το σημείο αυτό του ενιαίου μηχανισμού να βελτιωθεί με αλλαγή τη συνθήκη. Να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο. Νομίζω ότι το μήνυμα που λάβαμε από την ανταλλαγή αυτή απόψεων είναι ότι και ο Επίτροπο αλλά και εμεί, ω βουλευτέ, κάνουμε τη δουλειά αυτή σε ό,τι αφορά την κρίση το, που ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Προσπαθούμε να περάσουμε τις αλλαγές αυτές, προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε, να καταστήσουμε πιο ασφαλές το σύστημα και νομίζω ότι ένα τμήμα των ερωτήσεων σας απευθύνεται στο κατά πόσον τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία στο μέλλον. Πάντα λέω ότι όταν ε, υποβάλουμε ένα νομοθέτημα, μας ρωτούν στα μέτρα, στα μέσα ενημέρωση πότε θα εφαρμοστεί. Το 2014, όχι, διευκρινίζω, αυτή είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο πρέπει να καθυστερήσουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Σας ευχαριστούμε.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 Okay, I'm going to make a start. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε γιατί βλέπω ότι έχει έρθει ο εισηγητή. Έχουμε και του δύο εισηγητέ μαζί μα, τουλάχιστον του πιο σημαντικού εξ αυτών. Αυτές, αυτοί που αποφάσισαν να έρθουν. που αποφάσισαν να έρθουν. Το επόμενο θέμα είναι η ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο κύριο Τέρο είναι ο εισηγητή. Θα σα δώσω λοιπόν το λόγο για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μετά θα πάρουν το λόγο και οι σκιώτες συζητητές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να ξεκινήσω τη συζήτηση για το ακαθόδες αυτό το θέμα. Το κοινοβούλιο αυτό έχει καθήκον να εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να παραμείνουμε σε γρήγορση σε ό,τι αφορά την ισορροπία αυτή. Και το ερώτημα είναι το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας στον τομέα αυτό. Η ασφάλιση περιλαμβάνει προϊόντα στα μέτρα των πολιτών που θα λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές ε, συνθήκες. Έχοντας αυτά υπόψη, το τοπικό, αν θέλετε, πλαίσιο θα μπορούσε να εξυπηρετεί καλύτερα την ε, αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όχι απαραίτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ενιαία προσέγγιση για όλους δεν είναι η καλύτερη δυνατή στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για τις διαφορετικές ε, προτάσεις. Ελπίζουμε η Ευρώπη να προβεί τουλάχιστον σε μια ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Και αυτό από μόνο του είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και πολλά τέτοια περιστατικά και ακόμα και παρόμοια τέτοια ατυχήματα είναι δύσκολα στη σύγκριση. Αν υπομονώ να ακούσω τους ε, εμπειρογνώμονες και τις δικές σας θέσεις. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν από πλευράς από εξονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπούμε και σε λίγο παραπάνω λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πράσινη βίβλο αυτή ξεκίνησε μια πρώτη απόπειρα να καλύψει τέσσερις τομείς σε ό,τι αφορά την ασφάλιση κατά εναντί φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, σε ό,τι αφορά λοιπόν και την σχετική αποζημίωση. Η προσέγγιση που ακολουθείται εδώ σίγουρα δεν ε, ταιριάζει σε όλα τα κρατημέλη εξίσου. Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν ένα διαρκή κίνδυνο και έναν οικονομικό κίνδυνο. Και γι' αυτό υπάρχουν ε, σε κάποια κρατημέλη ασφαλιστικά συστήματα τα οποία λειτουργούν η τελευταία παλήρια στην ε, Γερμανία, η τελευταία πλημμύρα, είχε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι καταστροφές από την πλημμύρες του προηγούμενου έτους οδήγησαν σε διαφορετική ασφάλιση κινδύνου. Οι επιχειρήσεις πρόβλεψαν να μην υπάρχουν ζημίες στον επιχειρηματικό κλάδο, ακόμα και σε μικρομισές επιχειρήσεις, ενώ τα νοικοκυριά που δεν είχαν φροντίσει επαρκώς σε μία μικρή οικομόπολη, ε, αναλήφθησαν ακόμα και πρωτοβουλίε πολιτών για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων. Αν θέλουμε να βρούμε λοιπόν ευρωπαϊκέ λύσει για τον κλάδο αυτό, θα πρέπει, θεωρώ, να φροντίσουμε να μην καταπνίξουμε και να μην παραλύσουμε την ίδια πρωτοβουλία των πολιτών. Με τι ίδιε πρωτοβουλίε. μπορούμε να πετύχουμε πιο πολλά από την, με την πλήρη κρατική πρόβλεψη για τέτοιου κινδύνου. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της πράσινης βίβλου. Να μην λάβουμε μέτρα τα οποία τελικά θα καταπνίξουν την ίδια πρωτοβουλία από πλευρά των πολιτών. Και πάλι να σας αναφέρω πρόσφατα περιστατικά σε ό,τι αφορά πλημμύρες στην ε, κοινότητα Ντέκεντα στον ε, Δούναβη, ένα τρίτο των ε, νοικοκυριών έκαναν ασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες. Το 2 τρίτο τα δύο τρίτα δεν έκανε τέτοια ασφάλεια. Αν προβλέψει πλήρω το κράτο πλέον, ακόμα και το 1 τρίτο που είχε κάνει τι ασφάλειε, δεν θα το κάνει αυτό στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν έτσι να προσέξουμε σε ό,τι αφορά την ίδια ευθύνη, την παράλυση ενδεχομένω τη ίδια ευθύνη και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πρόβλεψη ασφαλίσεων, ελάχιστων ασφαλίσεων κτλ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο που έχω να θίξω, γιατί η πράσινη βίβλος αναφέρει το ποσοστό του κοινωνικού προϊόντος στα διάφορες χώρες, ε, κατά πόσον αυτό πλήττεται σε ζημίες φυσικά στην Δανία και στη Λιθουανία. Προκλήθηκαν οι πιο μεγάλες καταστροφές λόγω ανεμοθύελας, αλλά σε περίπτωση σεισμών υπερισχύει η Ελλάδα και η Ιταλία, σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία και η Αυστρία. Οι κίνδυνοι δηλαδή που υπάρχουν κατανέμονται διαφορετικά ανά χώρα και γι' αυτό λοιπόν οι λύσεις που προσφέρουμε θα πρέπει να λάβουν υπόψη ακριβώς αυτές τις ιδιαιτερότητες. Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείες σε ό,τι αφορά τις ε, ζημίε, σε ό,τι αφορά τι φυσικέ καταστροφέ, σε ό,τι αφορά του πυρηνικού κινδύνου, σε ό,τι αφορά ε, αέριο, πετρέλαιο και τα δικαιώματα ενημέρωση των ε, θυμάτων, ανθρωπογενείς καταστροφές και ό,τι αφορά τις αποζημιώσει και τη σχετική ρύθμιση. Υπάρχουν παραπομπές ε, στην οδηγία για τις ε, έρευνες ό,τι αφορά τις ασφάλειες και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Δεν είναι κάτι το αυτόματο που μπορεί να προσαρμοστεί στην αγορά. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ευθύνη και ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνης από το κράτος για την αξιολόγηση του θέματος αυτού. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή την πράσινη βίβλο που αποτελεί, αν θέλετε, πρόδρομο της λευκής βίβλου, να την εξετάσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αφήσουμε κατά μέρο τα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κ. Μπαλντίνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να, να πράξω αυτή την ευκαιρία και να μιλήσω κρατικά, να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο και όλους τους υπόλοιπους που μας ε, έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε διερμηνία από τα Κροατικά. Ελπίζω. Να με ακούτε καλά λοιπόν, μάλιστα πολύ ωραία, με καταλαβαίνετε, χαίρομαι. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η πράσινη βίβλος αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα σημαντικό και καλό σημείο φετηρίας για την έκθεση αυτή η πράσινη βίβλο. Εξηγεί πω έχει τρέχουσα κατάσταση, προσφέρει κάποιες λύσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλιση έναντι καταστροφών. σε ό,τι αφορά την έκθεση, θα πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσει να λάβει ενημερωμένο πλέον μια σωστή απόφαση. Η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται ακριβώς στη διάσταση αυτή. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο της ενημέρωσης του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητηθεί σε ό,τι αφορά και την υποχρέωση ασφάλισης. Επίσης περιλαμβάνονται κάποιες ιδέες σε ό,τι αφορά κάποιες σωματικές ασφαλίσεις και την ασφάλιση οργανώσεων. Θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή συμβαστική λύση αυτό το έγγραφο σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του καταναλωτή, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Επίσης πιστεύω ότι η απαραίτητη ισορροπία θα πρέπει να εξευρεθεί για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. χωρί την, ασφάλ... την ε, ισορροπία αυτή δεν θα μπορέσει να σημειωθεί σωστή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And, uh, Ευχαριστώ. Θαυμάσια διερμηνή είχαμε γιατί έχουμε καταπληκτικούς διερμηνείς και καταλάβαμε απόλυτα όλα όσα μας είπατε. Ο κύριο Τόρβαλτ από του Φιλελεύθερου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πράσινη Βίβλο και τον εισηγητή μα για τα εισαγωγικά του σχόλια. Οι θεομηνίε και ανθρωπογενεί καταστροφέ είναι δυστυχώ πρόβλημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πιο, ενησυχη... πιο είναι η τάση τη... που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο, ότι έχουμε όλο και περισσότερε τέτοιε θεομηνίε και καταστροφέ. Ε, τα τεκμηριωμένα επιστημονικά πορίσματα ότι θα ενισχυθούν οι κλιματικές αλλαγές ε, μας ε, καθιστούν πιο επίγουν σε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, πριν να θέσουμε υποέλεγχο έλεγχο τις κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα, όπως και τις ασφαλίσεις. Το, η πράσινη βίβλος δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο και το καλοκαίρι είχαμε τεράστιες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, στην Αυστρία, την Τσεχία και τη Γερμανία κυρίως επισκέφθηκα το Μαγδεβούργο πριν, μερικούς μήνες μετά τις πλημμύρες και το μόνο που μπορώ να πω ότι οι καταστροφές ήταν λιγότερες με, ε, από τις επιθέσεις του, ε, του 1630. Δεν ήταν τόσο βαρές οι ζημίες, αλλά πέραν τούτου ήταν εκτεταμένες οι ζημίες και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα και η πατρίδα του Σιγητή και η δική μου πατρίδα έχουν πληγεί από ακραία ε, μετεωρολογικά ε, φαινόμενα. Έχουμε χιονοθύελες ε, και δυστυχώς και οι καλοκαιρινές πλημμύρες εμφανίζονται τακτικά και φαίνεται ότι συστηματικά ο κόσμος υποτιμά τον κίνδυνο να γίνει θύμα θεομηνιών. Φαίνεται ότι είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι θα οφείλαμε και λιγότερο απεσιόδοξοι από ό,τι θα έπρεπε σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Ε, οι ακραίες καιρικέ συνθήκες είναι ένα καινούριο φαινόμενο και λέμε ακραίες ε, και γι' αυτό απρόθυμα υποθυμούμε, υποτιμούμε τον κίνδυνο και φυσικά ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει τις διαστάσεις ε, και του κινδύνου αλλά και των ζημιών και αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το θέμα της ασφάλισης. Ε, προτείνεται και ένα υποχρεωτικό σύστημα ασφαλίσεων στην Πράσινη Βίβλο. Δεν πρόλαβα να εξετάσω τι προβλέπουν τα κράτη-μέλη στα εθνικά του συστήματα, αλλά η πρόταση αυτή θέτει πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα. Για παράδειγμα, ε, θα πρέπει οι Έλληνες να διασώζουν τους Γερμανούς για πλημμύρες στον Έλβα και με μεγάλη ενυπομονησία περιμένω την απάντηση των Γερμανών. Και παρόλο που έχει νόημα μια τέτοια πρόταση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την προσωπική ευθύνη αλλά και των εθνικών αρχών σχεδιασμού. Γιατί μερικές φορές σωστή ασφαλτόστρωση βοηθάει καλύτερα να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επιδεινωθεί το σύστημα το φαινόμενο των πλημμυρών. Οπότε και το κράτος έχει ευθύνε. Επίσης υπάρχουν διάφορες διαδικασίες ε, για παράδειγμα κάποια έργα που μπορεί να γίνουν αλλά αυτά ίσως μειώσουν την αντικειμενική αξία των, αντικει... των ακινήτων. Υπάρχει δυνατότητα προληπτικών μέτρων. Βέβαια κατά πόσο τα προληπτικά μέτρα, αν δεν ληφθούν τα προληπτικά μέτρα και αυξηθεί ο κίνδυνος, ε, ε, αυξηθούν οι ζημίες μετά τις πλημμύρες, ποιος θα φέρει ε, την ευθύνη και ποιος θα πρέπει να πληρώσει τις ζημίες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παράδειγμα των Ελλήνων που θα διασώσουν του Γερμανού σε περίπτωση θεομηνιών, είναι θέμα το ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μήπως θα πρέπει να περιοριστούμε σε εθνικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε όμω ότι πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, γι' αυτό και δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ήμουν ήδη αρκετά προκλητικό με τι παρατηρήσει μου. Περιμένω με ανυπομονησία τι προτάσει του Φιλανδού συναδέλφου και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, αν θέλει, και στη συνέχεια στα φιλανδικά. Καλό είναι να είμαστε από και από προκλητικοί για να γίνεται πιο συναρπαστική συζήτηση. Ο κύριο Γκίγκολτ από του πράσινου. Καταρχά, πάντα μου προκαλεί έκπληξη το τι μπορεί να θεωρήσει ένα Φιλανδό προκλητικό. Εν πάση περιπτώσει. Προκειμένου να προκαλέσετε ένα Γερμανό, θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω ποσοστό προκλητικότητα, αγαπητέ συνάδελφε. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε που ακούμε ακροατικά. Καλώ ορίσατε. Αν υπομονούμε και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σα. Επί τη ουσία όμω, δεν έχουμε διαμορφώσει στην ομάδα μια κοινή γραμμή θα πρέπει να πω ότι έχω κάποιες πολύ βασικές αμφιβολίες για το όλο ζήτημα. Αναφέρθηκε και από τον Μπέρνερ Λάγκε προηγουμένως. Για το θέμα αυτό υπάρχει ένας, ε, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ηθικό κίνδυνο, μεγάλο πρόβλημα το οποίο και προκύπτει. Επειδή αν υπάρχει, πόσο, αν θέλετε, περίπτωση έλλειψης ασφάλειας, πάντα υπάρχει η ισχυρή τάση, μια πολιτική κοινότητα να έρχεται και να διασώζει αυτούς που δεν έχουν πληρώσει την ασφάλειά τους. Το βλέπουμε αυτό συχνά στην Γερμανία, επειδή είναι εθνικέ στιγμές, οι στιγμές, αν θέλετε, μεγάλων φυσικών καταστροφών. Είναι ε, περιπτώσεις όπου ο κόσμος ε, συμπονά αυτούς που έχουν πληγεί. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση διάσωσης. Ε, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κίνητρο να κάνει κανείς ασφάλιση και κατά δεύτερον, όπως είπε ο Βέρνερ Λάγκερ, να φροντίσει προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε αλλαγές. Και μεταξύ, αν θέλετε, των ακραίων αυτών ε, λύσεων, της υποχρεωτικής ασφάλισης, για παράδειγμα, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά. Τη υποχρεωτικής διάσωσης ουσιαστικά εκ των υστέρων ή του να λέμε ότι είμαστε μια χώρα που συμπάσχει και δεν θέλουμε να επιβαρυνθούν υποχρεωτικά και υπερβολικά άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου ενδεχομένως θα είναι πολύ ακριβή ασφάλιση. Χρειαζόμαστε μια αλληλεγγύη είτε με την χρηματοδότηση ε, μοντέλων ασφάλισης ή προβλέποντας ε, φτηνά ασφάλιστρα για τις εταιρείες ασφάλισης, τα οποία τελικά τα πληρώνουν άλλοι. Ή μία τρίτη λύση να αποδεχτούμε ότι πάντα θα υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις διασώσεων όπου μπορούν να εμφανίζονται οι πολιτικοί στις κάμερες κάποια κρίσιμη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να βρούμε λύσεις σε κάθε περίπτωση. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένο δε ότι χρειάζεται μία λύση ενιαία που θα ταιριάζει σε όλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένο. Θα ήθελα να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χρειάζεται και δικαιολογείται από πλευρά επικουρικότητα. να υπάρχει μια τέτοια λύση ενιαία για όλου. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω πιστεί καθόλου. Και είναι δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην ανακοίνωση όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Υπάρχουν, υπάρχουν ιδέες για το πού θα μπορούσε να έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία η Ευρώπη, για παράδειγμα έρευνα, ε, εμπειρίες, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στρατηγική για τη συντονισμένη διαχείριση διασυνοριακών κινδύνων. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να μην υπάρχει ηθικός κίνδυνος μεταξύ των κρατών μελών. να σηκώνει φράγματα, δηλαδή ένα κράτος μέλος ε, για να χτυπήσει η πλημμύρα πιο πολύ το διπλανό κράτος μέλος μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας σε ό,τι αφορά το Ρήνο για παράδειγμα ε, και άλλα παραδείγματα. Νομίζω ότι η Ευρώπη χρειάζεται αν υπάρχει πτυχή ανταγωνιστικότητας. Αν κάποιες χώρες για παράδειγμα έχουν ε, ασφαλίσει τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και έχουν εσωτερικοποιήσει το κόστος αυτός και αυξάνεται και μεγεθύνεται η αγορά ενέργειας και εδώ τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Δεν πρόκειται φυσικά ούτε για φυσικές ούτε για ανθρωπογενείς καταστροφές. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στις εργασίες μας, τις οποίες ε, θα παρακολουθήσει ο συνάδελφο Ζαν Κουλμπεσές που δεν μπορέσει να παραβηθεί σήμερα, θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή αυτή την ενιαία και ομοιόμορφη λύση για όλους. Να δούμε που τίθεται θέμα επικουρικότητας σε μια τέτοια κοινή λύση και θα ήθελα πολύ πιο σαφείς εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πού αξιολογείται διαφορετικά η αξία, το επιθυμητό επίπεδο αλληλεγγύης και που δεν χρειάζεται και που δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχω ακόμα απόλυτα πιστή και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει επιπλέον εξηγήσεις. Κύριε Καμάλ, σας ευχαριστώ πολύ ε, μιλάω εξ ονόματος του Ashley Fox, ο οποίος είναι σκιώδης ηγητής του ECR, επομένως ε, μου ζήτησε να διαβάσω κάποιες από τις σημειώσεις του. Θα προσπαθήσω να το κάνω με ενδιαφέρον τρόπο χωρίς να είμαι προκλητικός. Μην ζητάτε ποτέ από Γερμανούς και Βρετανούς να είναι προκλητικοί. Ο κύριος Φόξ λοιπόν χαιρετίζει την πρόταση αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ανταποκριθεί στην ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράσινη όμως βίβλο βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία δεν τον βρίσκουν σύμφωνο, ιδίως να αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση. Ε, πέρα από τις πρακτικές ε, δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν, όπως για παράδειγμα τις ε, εκτιμήσεις, πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει πραγματικά μια υποχρεωτική ασφάλιση σε περίπτωση καταστροφών, όταν ορισμένες οικογένειες έχουν πολύ περιορισμένους πόρους πλέον. Επίσης, αναφέρεται σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκαναν ορισμένοι συνάδελφοι. Σε περίπτωση καταστροφής, όποιος έχει τα μέσα είναι ήδη λογικά ασφαλισμένος και θεωρεί ότι η υποχρεωτική ασφάλιση θα πρέπει ενδεχομένω να αποφασιστεί σε εθνικό μόνο Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι αναφέρονται σε συνεχεί πλημμύρε που έχουν γίνει σε συγκεκριμένε περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά ο κόσμο δεν συμμορφώνεται και συνεχίζει και κτίζει κατοικίε περιοχέ αυτέ. Εν τέλει, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία καταβάλουν το τίμημα για τι καταστροφέ και όχι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένω θεωρεί ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε τι συμβάσει ασφαλιστικέ προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα του καταναλωτέ, να ενημερώσουμε καλύτερα τον Ευρωπαίο πολίτη και να καταφέρουμε να προλάβουμε κάποιε από τι καταστροφέ. Να αφήσουμε όμω το πεδίο επιλογή ελεύθερο για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ε, Ο θέλει να επανέλθει. Εν συντομία. Ναι, κάτι ξέχασα. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης, να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελείωσε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης 30 Ιουνίου. Ίσως θα πρέπει να ληφθεί κάτι άλλο υπόψη, ιδιαίτερα με τα νομικά, σε ό,τι αφορά τα νομικά συντήματα που ανέκυψαν. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας σχολιάσει εν συντομία το θέμα αυτό. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή, γιατί δεν έχω διαβάσει την πράσινη βίβλο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Αλλά και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις για το πού, πού είναι το κενό, πού είναι αυτό το χάσμα που προσπαθούμε να γεμίσουμε. Υπάρχει αυτή η προσθεθέμενη αξία, γιατί εξ όσων καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιες καταστροφές που δεν είναι, δεν είναι ασφαλίσιμες, δεν μπορούν να ασφαλιστούν. Τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε με λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες και να απαντήσετε και στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ε, δεν ξέρω, πού είναι η προσθεθέμενη αξία γεμίζετε κάποιο κενό, πώς βελτιώνετε την αγορά όπως αναφέρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ναι, συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, ίσως λοιπόν να μην απαντήσω συστηματικά ε, για αυτά που ρωτήσατε, Λούκας Μπάρτολα, από την Γενική Διευθύνση Μάρκτ, σε ό,τι αφορά και το τμήμα ασφαλίσεων και συντάξεων. Η Πράσινη Βίβλος είναι έργο διαφόρων ε, γενικών διευθύνσεων από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ΕΚΦΙΝ και ούτω καθεξής. Μεταξύ άλλων, ε, τάξου, ΤΕΦΚΟ και άλλες γενικές διευθύνσεις συμμετείχαν στην κατάρτιση της Πράσινης Βίβλου. Προσπαθήσαμε σε κάποιο βαθμό να ευαισθητοποιήσουμε για ένα θέμα το οποίο καθίσατε όλο και πιο σημαντικό στην Ευρώπη. Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Στην Πράσινη Βίβλο, λοιπόν, προσπαθήσαμε να είμαστε κι εμείς λίγο προκλητικοί, αλλά και παιδαγωγικοί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, να κατανοήσουμε κατά πόσον η Ένωση μπορεί να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν βρει κάποιες λύσεις, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις φυσικές αλλά και τις ανθρωπογενείς καταστροφές, αλλά και υπάρχουν και πολλά κρατημέλη που υστερούν στο σημείο αυτό. Άρα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα αυτό και να μάθουμε ημένα από τους δε. Ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών, αλλά θέλουμε επίσης να κατανοήσουμε κατά πόσον οποιαδήποτε δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νόημα στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία διαβούλευσης. Μέχρι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, οι Λάβαμε 65 απαντήσεις από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, από εθνικά κοινοβούλια, κυβερνήσεις, καταναλωτές και ασφαλιστικές, τις οποίες και αξιολογούμε στην παρούσα φάση οι απαντήσεις αυτές θα δημοσιευτούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας, όπως και η σχετική αξιολόγησή μας. Ευχαριστώ. 65. 65 απαντήσεις λάβατε στη διαδικασία διαβολούς. 75. Και τι είδους οργανώσεις έστειλαν τις απαντήσεις τους. Αν θυμάμαι καλά, από εταιρείε ασφάλισης, αντασφάλισης, ενός εταιρεών ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και τοπικές ή εθνικές βουλές, κυβερνήσεις και οργανώσεις καταναλωτών. Δεν ξέρω αν απαντήθηκαν τα ερωτήματά σας. Ίσως ε, τις απορίες μας θα μπορούσαμε να σας τις στείλουμε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αυτός ο τρόπος που συνήθως ε, αντιμετωπίζουμε τα θέματα, αλλά η πολιτική είναι απρόβλητη μερικές φορές. Δεν θέλουμε πρώτη φορά να σας τριμώξουμε. Τώρα ο εισηγητής μας πώς ε, θα συνεχίσει, πώς θα συνεχίσει με την ε, παρουσίαση της έκθεσής του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδέλφων και βλέπω ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύγκληση απόψεων. Οπότε μπορώ να συνεχίσω την εκπόνηση της έκθεσης και στο κείμενό μου σκοπεύω να λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Σίγουρα θα καταλήξουμε σε μια έκθεση που απελπιστώ ότι θα τύχει ευρεία ε, αποδοχή. Στι 14 ε, Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. Ελπίζω να έχουμε πρόσβαση στι διαβουλεύσει, να γίνονται ηλεκτρονικά. 22 Οκτωβρίου λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες, θα τις εξετάσουμε 25-26 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 17 Νοεμβρίου, προκειμένου να περάσει η έκθεση αυτή στην πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρέμβαση και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Yeah, so we, we're a little bit of, we're a little bit ahead of schedule. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα την προηγούμενη έκθεση, 10 λεπτά νωρίτερα. Γι' αυτό και περιμένουμε τον κύριο Μπερτό. Α του τηλεφωνήσει κάποιο να δούμε μήπως είναι στο δρόμο ήδη. Okay, well, we have... δεν απαντά στο γραφείο. Καλά, τότε θα τον περιμένουμε. Um, yes. We have our shadows here. Οι σκιώδεις μας ηγητές πάντως είναι παρόντες. Ένας τουλάχιστον, η κυρία Μία, η κυρία Κλέβα. Ούτε ο Σβέν. Α, όχι, εκεί είναι. Απλώς μετακόμισε. Αλλού κοιτούσα. Και ο Σβέν είναι εδώ. Έχουμε δύο σκιώδης Μας λείπουν ο εισηγητή της γνωμοδότησης και ένας σκιώδη Ο λιγόλεπτη διακοπή, αλλά παρακαλώ μην φύγετε. μη μου τη σκάσετε. Γιατί μετά που να σα ξαναβρούμε. Είμαστε καλά στην ώρα μας σήμερα. Ελπίζω να τελειώσουμε και λίγο νωρίτερα. Παρακαλώ να τηλεφώνουμε εγκαίρως τους συζητητές. Να. να καλέσουμε και τον μεθεπόμενο. Α, δεν έχουμε άλλο θέμα μετά του κυρίου Μπερτό. Non, oui, oui, euh, on attend M. pour la prochaine rapport. Parce qu'on a, on a un peu... On a... Περιμένουμε τον κύριο Μπερτό, γιατί τελειώσαμε νωρίτερα, πέντε λεπτά νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Επομένω, αναμένουμε τον κύριο Μπερτό για να καλύψουμε το τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Les, les shadows sont là. όμως ηγητές είναι ήδη εδώ. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο εισηγητής έχει καταφτάσει. Και όπως πάντα λέω, εδώ είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι. Οι σκιώδεις, αυτοί που θα εργαστούν για το θέμα αυτό. αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί. Ο κύριος Μπέτο, αν θα μπορούσατε παρακαλώ να κάθετε. Sorry. Je ne parle pas italien. Δεν θα μιλήσω τελικά. Γερμανικά, μάλιστα. Γαλλικά, ναι. Και λίγα τουρκικά. Μέχρι εδώ όμως. You're leaving, but you're one of my shadows. Don't leave. Μα είστε σκιώδε, μην φύγετε, σας παρακαλώ. Oui, c'est ça. Um, Καλώς ορίσατε. Συγγνώμη, αλλά τελειώσαμε λίγο πιο νωρίς το προηγούμενο θέμα, γι' αυτό σας περιμέναμε. Δεν καθυστερήσαμε και με την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και πάντα είναι ενδεικτική η ώρα ασφαλώς. Το υπενθυμίζω αυτό πάντα. Ε, χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και σας δίνουμε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς ε, σας ζητώ συγγνώμη για τα όσα θα πω στην συνέχεια. Πρώτη φορά παρουσιάζω ως Ευρωβουλευτής ε, μια εργασία μου εδώ πέρα στην Επιτροπή, επομένως συγγνώμη για ενδεχόμενα λάθη που θα κάνω. Θα ήθελα Όχι, όχι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή απλώ τελειώσαμε λίγο νωρίτερα. Λογικά θα πρέπει να περιμένετε, δεν θα είχαμε αρχίσει την ώρα μα. Απλώ ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε. Σε κάθε περίπτωση ενδεχομένω να έχω κάνει όμω και λάθη στο ίδιο το κείμενο το οποίο έχω συντάξει. Όσον αφορά τώρα το θέμα αυτό το οποίο μου ζητήθηκε να αναλύσω και να επεξεργαστώ, δηλαδή την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα εταιρικά έσοδα, Προσπάθησα να αξιολογήσω τους τρόπους, τα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ουσιαστικά σκέφτηκα ορισμένα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να προτείνουμε στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Από τη μια θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια συμμετοχή των εργαζομένων στη χρηματοδότηση της εταιρεία μέσω της συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο ή μέσω ειδικών πιστοτικών τίτλων, δηλαδή μέσω ομολόγων ομολόγων της εταιρείας αυτής στην οποία εργάζονται. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό καθεστώς δεν θα έχει να κάνει με την ίδια την εταιρεία, αλλά μπορεί να βαρύνει τους ίδιους εργαζομένους με βάση το ποσό αυτό το οποίο θα μπορούσαν να λάβουν ως αποδοχή και ενδεχομένω να προβλεφθεί μια φορολογική διευκόλυνση γι' αυτό. Μια άλλη μορφή χρηματοδότησης, συμμετοχής δηλαδή των εργαζομένων σε εταιρικά έσοδα θα ήταν να υπάρχει ένα μέρος της αμοιβή το οποίο θα καταβάλλεται μέσω μετοχών, μέσω τίτλων δηλαδή της ίδιας της εταιρεία που θα εκδίδονται ειδικά για τους εργαζομένους ή μέσω των κλασικών μετοχών της εταιρεία αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να είχαμε μια φορολογία υπέρ της εταιρείας αυτής προσπαθώντας ουσιαστικά να συγκλίνουμε λίγο περισσότερο αυτό το οποίο δίδεται ως αμοιβή στον εργαζόμενο με την πραγματική αντικειμενική αξία της μετοχής αυτής. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η ε, ονομαστική αξία αυτού του τίτλου, η αγοραία αξία αυτού του ομολόγου, η λογιστική αξία στις οικονομικές καταστάσεις εταιρεία. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το φορολογικό καθεστώς το οποίο θα ισχύει για αυτές τις εταιρείε, οι οποίες αποφασίζουν κατά αυτόν τον τρόπο να επιμερίσουν τα κέρδη τους ε, στους εργαζομένους τους. Ένα άλλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρεία τους θα μπορούσε ιδίω στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης να είναι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε μία συμμετοχή μέσω συνεισφορών των εργαζομένων, πρώην εργαζομένων, οι οποίοι δηλαδή έχουν απολυθεί από την εταιρεία εξαιτία της οικονομικής κρίσης ή μιας κρίσης τη ίδια εταιρείας. Θα μπορούσαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μέσω των αποταμιεύσεών τους ή μέσω των επιδομάτων ανεργίας τους, να χρηματοδοτήσουν ε, την ανάκαμψη της εταιρεία αυτής ή να χρηματοδοτήσουν ε, περαιτέρω δραστηριότητες ή επενδύσεις εταιρεία αυτής με απότερο όμως στόχο την ε, επαναπασχόληση των ε, εν λόγω πρώην εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας του κινδύνου όσον αφορά αυτού του είδους χρηματοδότησης των εταιριών και νομίζω ότι η οίκη αξιολόγησης ε, πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει ή τουλάχιστον κάποιοι άλλοι οργανισμοί πιστοτικοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με την έκδοση αυτών των τίτλων να αναλύσουν όλους τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με αυτού του είδους την ε, επένδυση και με αυτού του είδους τη χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά πρότυπα όσον αφορά τις εταιρείες οι οποίες είναι συγμένες στο χρηματιστήριο και τις εταιρείες εκείνες οι οποίες δεν είναι συγμένες στο χρηματιστήριο, δηλαδή συνήθως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι η μετοχή μιας εταιρείας η οποία είναι συγμένη στο χρηματιστήριο μπορεί άμεσα να, ε, να, να δοθεί, να αγοραστεί ή να ασχοληθεί. Επομένως, ανήκει σε, μια ξεχωριστή, σε ένα ξεχωριστό νομοθετικό καθεστώς. Αυτά είχα να πω όσον αφορά το περιεχόμενο της γνωμοδότησής μου και είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για περαιτέρω ερωτήσεις. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για συγκεκριμένες πτυχέ γνωμοδότησης και για τι υπόλοιπε πτυχέ αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόληση. Να ακούσουμε τους Κιώδης τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά κάποιου τομεί τη γνωμοδότησης αυτή, γιατί μιλάμε για φορολογικά κίνητρα, υπερβολικού κινδύνου στον επιχειρηματικό κλάδο και προκλήσεις που αφορούν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Είναι δική μα η κλάδη αυτή και νομίζω ότι έχουμε πλήρη αρμοδιότητα. Να ακούσουμε τους Κιώδης που συμμετέχουν στην ομάδα και θα σας βοηθήσουν στην γνωμοδότηση αυτή. Κυρία Κλίδα, καταρχά στο κατάλογο μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερτότ, τον εισηγητή μας, για τη συνεισφορά του στην πολύ αυτή σημαντική συζήτηση για την οικονομική συμμετοχή των ε, εργαζομένων στις εταιρείε. Τα πρόσφατα τελευταία χρόνια η όξυνση της κρίσης ε, και ο μεγάλος αριθμός ε, των πτωχεύσεων, αφαιρεγγιότητας, των επιχειρήσεων και των κρατικών και των ιδιωτικών ε, ανέδειξαν την ε, ανάγκη διαφόρων μορφών συμμετοχής ε, των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Και άλλο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι η τάση αυτή υποστηρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό τώρα πλαίσιο για να καθορίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές τέτοιων πλαισίων και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε την αμοιβαία αναγνώριση τέτοιων ε, συστημάτων συμμετοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να προτείνει ένα ομοιόμορφο νομικά πλαίσιο για την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων και ο Επίτροπος Μπαρνέ ήδη ε, είχε κάνει την υπόσχεση αυτή σε μια περσινή δημόσια κρόση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πιο μακρό πρόθεσμο όραμα και μια βιώσιμη συμμετοχή και επίση να είναι οικειοθελή προαιρετική αυτή η βάση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να αφήσουμε τη διακριτική ευχαίρεια στου εργαζόμενου για το κατά πόσο θα συμμετέχουν ή όχι σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα φορολογικά κίνητρα και οι σχέσει με τη μισθολογική πολιτική ή τη συμμετοχή στα κέρδη, θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να υποβάλλονται στους εργοδότες, στου και τα συνδικάτα. Επίση, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε τις βέλτιστες πρακτικές και τα καλύτερα ευρωπαϊκά υποδείγματα να τα να γνωστοποιήσουμε σε όλη την Ευρώπη γιατί σίγουρα η κατάσταση είναι διαφορετική στο Βορρά και στο Νότο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ε, την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Επίσης, τα φορολογικά ζητήματα είναι τα πιο σημαντικά. Το πρόβλημα της πιθανή ε, πιθανής διπλής φορολόγησης που θα περιορίσει πολύ σοβαρά την ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, εθνικές αρχές ε, στη χάραξη και πρόταση για τις φορολογικές διευκολύνσεις και τα φορολογικά κίνητρα που μερικές φορές είναι το κλειδί για την επιτυχή συμμετοχή των εργαζομένων στο σύστημα. Επίσης, ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους ε, σε μετοχές, θα πρέπει και εκεί να δούμε ποια, σχέση θα έχει με τις επενδύσεις στα συνταξιδοτικά συστήματα και επίσης ποιο μερίδιο θα αφαιθεί σε αυτή την συμμετοχή στις μετοχές. Επίσης δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στις εταιρείε να αντικαταστήσουν τους, τα συστήματα κερδών από τη συμμετοχή των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είναι νέο το πλαίσιο και είναι σημαντική μακροπρόθεσμη στόχη και να είναι προαιρετική η βάση. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην αρχή της ισότητας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν και να δίνονται να ε, συμμετέχουν στο σύστημα. Επίσης θα πρέπει η αρχή της επιμέλειας ε, να ληφθεί υπόψη, δηλαδή όλοι οι ενεχόμενοι να επιδεικνύουν την απαραίτητη ε, φρόνηση, σοφροσύνη, επιμέλεια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την γνωμοδότηση και προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμπάκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ καταρχά τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Θεωρώ ότι όλη η συζήτηση επικεντρώνεται με την, έχει να κάνει με τη συζήτηση που έχει να κάνει με την διαχείριση των ε, εταιριών. Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη αυτό, γιατί ασφαλώς αυτό δεν αφορά μόνο θέματα αμοιβή. Άρα, κοιτάμε το θέμα αυτό της αμοιβή, της συμμετοχής των ε, υπαλλήλων και σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή για τον κίνδυνο και θα πρέπει να, να εξασφαλίσουμε ότι, ότι όλα τα κίνητρα που δίδονται και για τους υπαλλήλους αλλά και για τι ε, τις επιχειρήσεις είναι ίσα. Και νομίζω ότι με τα συστήματα αυτά το πετυχαίνουμε αυτό. Φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι θελούσιο, θα πρέπει να προσφερθεί κάποια στιγμή στους ε, υπαλλήλου που θέλουν να συμμετάσχουν. Και στη δική μου χώρα να σας πω ότι δεν είναι πολύ ίσως αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που ενέχει και κάποιο κίνδυνο ασφαλώς. Η οικονομική συμμετοχή λοιπόν σε μια επιχείρηση μπορεί να πάει καλά, μπορεί και όχι. Άρα οι πληροφορίες που παρέχονται στους υπαλλήλους είναι θεωρώ κρίσιμη σημασίας σχετικά με τον κίνδυνο που ελοχεύει. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον θα πρέπει να συμμετέχουν και οι και αξιολόγηση, ε, γιατί, όπως είπατε, πρόκειται για, ένα, για μια ρευστή αξία για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Για τις μικρομεσαίες όμως δεν είναι ρευστή αυτή η αξία. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κίνητρα στις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί προσθήκη στην αμοιβή των υπαλλήλων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το μισθό ενός, ούτε ποσοστιά, ούτε πλήρως το μισθό ενός ατόμου. Επίσης και η φορολόγηση θα πρέπει να είναι διαφορετική. Άρα και η διπλή φορολόγηση σε εντεσνοριακό επίπεδο θα πρέπει να εξεταστεί, αλλά και η εναρμόνιση γενικότερα σε θέματα φορολόγησης μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, προτείνεται όλοι οι υπάλληλοι να έχουν δυνατότητα να μπορούν να επανεπενδύουν τα κεφαλαία τους στις εταιρείε. Αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Είναι ίδιοι όροι όπως και για τους εξωτερικούς επενδυτές. Γιατί να υπάρχει διάκριση λοιπόν μεταξύ των πρώην υπαλλήλων που είναι συνταξιβετημένων για παράδειγμα των εξωτερικών επενδυτών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ίση αντιμετώπιση. Άρα και εμείς θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες τροπολογίες, αλλά θεωρώ καταρχάς ότι είναι σημαντικό το θέμα της αμοιβή και της επιπρόσθετης αμοιβή των ε, υπαλλήλων. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ ευρύτερα, γιατί θεωρώ ότι δίνει καλή κίνητρα στην ε, επιχείρηση προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του οράματο, αν θέλετε, και τη πράξη τη επιχειρήση. Μάλιστα, να επανέλθουμε λοιπόν στον εισηγητή, γιατί δεν είναι εδώ πέρα ο Σκιώδη από του πράσινου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις που κάνανε, για το ότι τόνισαν μια πτυχή την οποία εγώ δεν είχα τονίσει αρκετά στο γνωμοδότησή μου και η οποία όμως αναφέρεται. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην εθελοντική βάση που θα πρέπει να έχει το σύστημα αυτό. Στην πρώτη μάλιστα παράγραφο αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στο ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να είναι εθελοντική από τους απασχολούμενους. Και μάλιστα κλείνω την παράγραφο αυτή λέγοντας ότι ε, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιοδήποτε μέτρο έχει να κάνει με την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα τερικά έσοδα θα πρέπει να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα και μάλιστα θα πρέπει να γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση. Λέω επίσης ότι ε, θέλω να είναι σε θέση οι απασχολούμενοι να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Κατά αυτόν τον τρόπο οι απασχολούμενοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή μέσω εξωτικών ταμείων που έχουν ιδρυθεί ιδιωτικά μπορούν να συμμετέχουν και κατά αυτόν τον τρόπο στα εταιρικά έσοδα της εταιρεία. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουν ένα μεγαλύτερο μέγεθος και βαρύνουν περισσότερο, αν θέλετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας όσον αφορά το ότι πρέπει να ομογενοποιήσουμε τη συμμετοχή, τις επενδύσεις των πρώην απασχολούμενων, των απασχολούμενων ή οποιονδήποτε εξωτερικών επενδυτών. Εγώ θεώρησα ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να τονίσουμε απλώς την δυνατότητα των πρώην εργαζομένων, και όταν λέω πρώην εργαζόμενοι δεν εννοώ αυτούς οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους κύκλο, αυτούς δηλαδή που συνταξιδοτήθηκαν. Αναφέρομαι σε πρώην εργαζόμενους οι οποίοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την εταιρεία και οι οποίοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κάποιες νέες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επαναπασχόλησή τους. Είπα ότι αυτή η επαναπασχόληση θα πρέπει σε πρώτο βαθμό να αφορά τους ίδιους που έχουν απολυθεί και στη συνέχεια ενδεχομένω και άλλους. Ενδεχομένως η διάταξη αυτή να μπορεί να βελτιωθεί αποτελεί πάντως λεπτομέρεια στα πλαίσια μιας πιο γενικής διάταξης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καλή αυτή η γνωμοδότηση και πολλά θετικά σχόλια ακούσαμε από τους ε, σκιώδεις. 30 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογίων. Στις 25 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η ψηφοφορία. Στην Ολομέλεια θα περάσει αυτό μετά από την έγκριση φυσικά της Επιτροπής Απασχόληση στις 13 Ιανουαρίου. Να σας υπενθυμίσω στους τελευταίους αναπομείνοντες εδώ που μείνατε μέχρι τέλους. Αύριο το πρωί ξεκινάμε στις 10, όχι στις 9. Η ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τους εκπροσώπους των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων έχει προγραμματιστεί από τις 3 μέχρι τις 4.30 αύριο το απόγευμα και δεν έχουμε τίποτε άλλο μετά, μετά τις 4.30, μετά τις συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα πολύ θετικά σας σχόλια.